<coughs> Αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, θα αρχίσει η συνεδρίαση μα τώρα. Καταρχήν κάποιε προαναγγελίε. Φιναδικά, φιλολογικά και λιτοδανικά, ουγγαρικά δεν προσφέρονται σήμερα. Έχετε τη πλησία διάταξη μπροστά σα, δεν υπάρχουν παρατηρήσει από ε, Θεωρείται λοιπόν εγκεκριμένη η ημερησία διάταξη. It's now, now it's, it's Εντάξει τώρα, ωραία. Αυτή η συνεδρία μεταβιβάζεται σήμερα, ζωντανή αναμετάδοση. Στις 9 Φεβρουαρίου 2009 με την ΑΦΕΤ θα έχουμε ένα ε, εργαστήριο για το θέμα της ασφάλειας. Προβλέπεται να ε, ολοκληρωθεί αυτή η συνεδρίαση με μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Πριν από τα τέλη της αιτίας πρέπει να κάνουμε κάποια δήλωση όσον αφορά το θέμα της security. Η συνάδελφος Ιστάντε επέμεινε πάνω σε αυτό ιδιαίτερα. Είναι καλή η δυνατότητα αυτή νομίζω που έχουμε μετά από μια συζήτηση του θέματος να προετοιμάσουμε ενδεχομένως και ένα ψήφισμα. 10 Φεβρουαρίου 2009. Πρόταση της σύστασης της κυρίας Μπέρ όσον αφορά την σύμβαση μη διάδοσης ε, πυρηνικών όπλων. Κύριε Βενέρα, προσωπική εκπρόσωπος του κυρίου Σολάνη για αυτό το θέμα, ελπίζουμε να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση. Όσον αφορά τώρα το θέμα της σημερινής μας ε, συνεδρίαση, θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και το θέμα της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής ασφάλειας. Ε, σε αυτό το κείμενο η τρομοκρατία απαριθμάται σαν μια από τις κύριες απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτού έχω τον συντονιστή της αντιτρομοκρατικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζιλ Κερκόβε, και επίσης δύο εκπροσώπους της Interpol, τον κύριο Πιέρ Μπολάντ, ειδικό εκπρόσωπο της Interpol στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον κύριο Βασίλειο Θεοφιλόπουλο, ειδικό αξιωματικό σε θέματα τρομοκρατίας και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω του συναδέλφου τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που έχουν εκκληθεί να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή. Όπω σα είπα, η τρομοκρατία είναι με κύριε απειλέ των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Η καταπολέμηση της βασίζεται καταρχήν στη συλλογή πληροφοριών που δίνουν τη δυνατότητα να ε, αποτραπεί η τρομοκρατική απειλή πριν δράσουν οι τρομοκράτες. Και γι' αυτό η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απολύτως απαραίτητη μεταξύ όλων των υπηρεσιών που έχουν πληροφορίες για ε, τρομοκρατικά δίκτυα. Η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων αυτών και των θεσμικών οργάνων όπως Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, Ιντερπολ και μεμονωμένων κρατών θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και τα κράτη μας από την τρομοκρατική απειλή. Γι' αυτό στην ίδια συνεδρίαση έχω καλέσει το συντονιστή Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπροσώπου της Ιντερπολ για να μας εξηγήσουν πώς συνεργάζονται οι δύο αυτές οργανώσεις και πώς ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τους. Θα ήθελα να ξέρω επίσης πώς συλλέγουν οι πληροφορίες και τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιντερπολ και άλλες οργανώσεις για να θέσουν εκτός μάχης και να καταστρέψουν τον νομοκρατικά δίκαιο. Ο κύριος Δεκέρκοφ έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Νομίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας. Μου δώσατε ένα δεκάλεπτο τέταρτο. Θα προσπαθήσω λοιπόν σύντομα και συνοπτικά να σας αναφέρω τα βασικά στοιχεία της έκθεσης που παρουσίασα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως επίσης να σας αναφέρω και πώς λειτουργεί το σύστημα ανταλλαγών πληροφοριών με την Interpol. Εγώ σας έδιδωσα έναν απολογισμό του τελευταίου εξαμήνου που δίνει μια συνοπτική εικόνα για τις σχέσεις μας με την Interpol και για το τι κάνουμε. Το πρώτο σημείο, το βασικό, είναι η ανταλλαγή πληροφόρησης. Και διακόπτεται το μικρόφωνο του ομιλητή, δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, εμείς εργαστήκαμε σκληρά από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά και ακόμη περισσότερο μετά τις τρομοκρατικές ε, δράσεις στην ε, Μαδρίτη ε, για το θέμα της ανταλλαγής δηλαδή πληροφοριών σε αστυνομικό επίπεδο. Και έχουμε θέσει σε δίκτυο τις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών, ε, τις τράπεζες δεδομένων για τα δακτυλικά αποτυπώματα και το ADN. Έχουμε φτιάξει μια τράπεζα αρκετά επεξεργασμένη τράπεζα για τα χαμένα και κλεμμένα διαβατήρια και θα έχουμε σε κάποια φάση τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε παντού στην επικράτεια στα σύνορα αν κάποιος έχει στην κατοχή του ένα διαβατήριο κλεμμένο ή χαμένο. Εκεί που θα επιμείνω και όπου θα παίξει σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο είναι ο καθορισμός μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το πώς συλλέγεται και το πώς μετά ε, ανταλλάσσεται η πληροφορία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα γενικότερο όραμα για το τι θέλουμε να κάνουμε ως προς τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφόρησης. Λείπει λοιπόν ένα όραμα, όπως και λείπει, λείπει επίσης και ο καθορισμός των ορίων. Εμείς δεν θέλουμε να συλλέγουμε στοιχεία για όλο τον κόσμο οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς θέλουμε να περιορίσουμε τη συλλογή πληροφοριών σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο, διότι εμείς έχουμε ως αρχή να προστατεύουμε τα ατομικά προσωπικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν εμείς να διαπιστώσουμε καταρχήν ποιες είναι οι ανάγκες μας και δεύτερο, μέσα σε μία πολιτική και στρατηγική οπτική να θέσουμε τα όρια μας. Και για το θέμα της διάθεσης των ε, στοιχείων, αλλά και για να διασφαλίσουμε τους συμπολίτε μας. Υπάρχουν και άλλα ε, σχέδια, τα, ε, τα οποία βρίσκονται στα σκαριά, Έχουμε την απόφαση του 2005 που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να τροφοδοτούν και την Europol και την Eurojust με πληροφορίες και για τις ε, έρευνες αλλά και για τις διώξεις. Επίσης, ε, ε, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το ε, το Czech Web Europol, αυτό που έτσι το ονόμασαν οι Γερμανοί, δηλαδή να βάλουμε μαζί όλα τα στοιχεία που έχουμε στις έρευνες που γίνονται σε επίπεδο ίντερνετ. Προσπαθούμε λοιπόν να θέσουμε σε κοινή βάση όλες μας τις πηγές. Επίσης, μετά από την ανταλλαγή των πληροφοριών, είναι αυτό το τεράστιο πεδίο της πρόληψης. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα λεπτό από πολιτικής πλευράς, είναι ιδιαίτερα ε, δύσκολο να καθορίσει κανείς ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν κάποιο, ένα άτομο στον εξτρεμισμό. Προσπαθώ λοιπόν να δω πώς λειτουργεί αυτή η νέα προσέγγιση και τι αποτέλεσμα δίνει. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε τα κράτη που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία και που θέλουν να αναλάβουν ένα ρόλο leadership, ένα ρόλο αρχηγικό στον τομέα αυτό. Εγώ διαπίστωσα ότι τέτοια κράτη είναι έξι και καταφέραμε μαζί με τους Βέλγους δηλαδή εχθές να βρούμε 7 κράτη. Και προσπαθούμε να συλλέξουμε τις καλύτερες πρακτικές και να τις διαδώσουμε στα κράτη-μέλη. Δηλαδή πώς παρακολουθούμε την διάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ε, αστυνομία εγκύτητας, δηλαδή το πώς λειτουργεί η τοπική αστυνομία στη συλλογή της πληροφόρησης, αλλά και στη διαπίστωση ε, ρίζοσπαστικών ε, θέσεων. Και συμμετείχα μάλιστα και σε ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και πίστηκα ότι το θέμα της πρόληψης είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί σε επίπεδο τοπικό. Με την Ολλανδία συνεργαζόμαστε στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Και μετά θα σας μιλήσω και για τον Κουαντάναμο. Η Ισπανία αποφάσισε να εργαστεί στο θέμα της κατάρτισης των ημάμιδων διότι υπάρχει μία διαφορά στο πώς ε, καταρτίζονται αυτοί οι ιερωμένοι διότι υπάρχουν κράτη όπου όπου ο διαχωρισμός ε, θρησκείας και κράτου είναι σαφέστατος, παράδειγμα η Γαλλία, που καταρτίζει επιμορφώνει τους ημάμιδες για το πώς θα διαχειριστούν ένα τζαμί ή για το πώς θα δουλέψουν ως σύμβουλοι στις φυλακές. Επίσης θέλουμε να ορίσουμε το how to counter the single narrative, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν αντίλογο. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε εμείς να διατυπώσουμε έναν αντίλογο στο λόγο που προφέρει η Αλκάιντα για το Πακιστάν, για το Αφγανιστάν, αλλά και για το Μαγκρέμπ. Είναι πάρα πολύ εξεζητημένος ο λόγος της Αλκάιντα, αυτά τα οποία προφέρει ως θεωρία. Με τους Γερμανούς εμείς συνεργαστήκαμε και διαπιστώσαμε την τεράστια δύναμη που έχει η Αλκάιντα στην περιοχή και το πώς κινητοποιεί μέσα από βίντεο, μέσα από το ίντερνετ και γενικά μέσα από, την, ε, από τα συστήματα επικοινωνίας. Θεωρώ ότι σε αυτή τη μάχη των μίντια πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα οι δημοσκοπήσεις στον αραβικό κόσμο και πριν ε, ε, παρέμβει το Ισραήλ στη Γάζα δίνουν ότι η αρχίζει και πέφτει η υποστήριξη του μουσουλμανικού κόσμου για την αλκαΐδα τον, ε, και τον Μπι Και αν δείτε το YouTube και δείτε και τα βίντεο που βάζουν στο YouTube οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά φιλμάκια τα οποία είναι κατά του Μπιν Λάντεν. Εγώ έχω υπόψη μου δε και τον δόκτορα Ελφάντελ Ολίβ ο οποίος ε, προσπαθεί να ενισχύσει τους ε, μετροϊοπαθείς ε, μουσουλμάνους να αντιπαρατεθούν στο ριζοσπαστικό Ισλάν. Πάμε τώρα στην εξωτερική διάσταση που είναι πάρα τώρα, πολύ σημαντική για αυτή την Επιτροπή. Τώρα όμως δεν έχω πολύ χρόνο να αναπτύξω τα θέματα αυτά, αλλά θα προσπαθήσω εν το μέτρο του δυνατού να είμαι παρόν και να βοηθήσω τους συναδέλφους να μπορέσουν να καταρτήσουν μία συνολική στρατηγική σχετικά με τις δύο βασικές επιπρόσθετες προτεραιότητες μας, το Πακιστάν ε, και ε, τη τις, ε, τις ε, περιοχές και το Σαχέλ όπου ξέρετε ότι ε, είναι οι δύο πιο επικίνδυνες περιοχές. Ξέρετε στο Σαχέλ η Αλκάιντα είναι πάρα πολύ ενεργή, ενδιαφέρεται, έχουν πολλά συμφέροντα στο Μαγκρέβ και ε, το βασικό θέμα είναι η σχέση με την Ευρώπη και η άμεση στήριξη την οποία μπορεί να έχει οργάνωση αυτή στην Ευρώπη. Ε, επιπλέον αντιμετωπίζουμε ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών τα οποία μεταφέρονται προς την Ευρώπη, ξεκινάνε από τη Γουινέα Βισάου, προχωράνε προς τη Μαυριτανία και από εκεί περαιτέρω. Συγχρόνως ε, λαθρεμπόριο ε, από ε, πλαστά εμπορεύματα, από εμπόριο ανθρώπων και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή διάφορα θέματα τα οποία ε, ενδιαφέρουν τους ε, Ευρωπαίους και γι' αυτό προσπαθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξουμε από τη μία μεριά την ασφάλεια και από την άλλη μεριά την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία χωρίς να εξετάσουμε γενικότερα την ασφάλεια και ξέρουμε ότι το θέμα είναι πολύ βασικό και είναι πολύ πιο σημαντικό και υπάρχουν πολλά περισσότερα, ε, περισσότεροι ευρωβουλευτές οι οποίοι κοιτάνε πώς μπορούμε να τονίσουμε την ε, πολιτική πτυχή για να αποφύγουμε την τρομοκρατία. Και ε, με το Πακιστάν πρέπει να εξετάσουμε ε, την προθυμία της, του Πακιστάν να συμπράξει μαζί μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πόσο μπορούμε να εξετάσουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Μουμπάι έκανα μία επίσκεψη η οποία ε, επιβεβαίωσε την ανάγκη ότι πρέπει να βοηθήσουμε το Πακιστάν διότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας όχι μόνο στη δυτική πλευρά δηλαδή κοντά στο Αφγανιστάν δηλαδή εκεί που έχετε ε, μία τεράστια αναταραχή ε, διότι είναι η ΣΥΑ εναντίον των Σούνι και ακόμη πιο προβληματικά στο Πουντζάμπ υπάρχει η μία ε, τρομοκρατική ομάδα, η JUD, η οποία είναι πολύ πιο προηγμένη και στενά συνδεδεμένη με την Αλκάιντα και δραστηριοποιείται στην Ινδία και στο Μουμπάι. Αυτό που απεκόμισα από την επίσκεψη αυτή είναι η σημασία που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πακιστάν διότι έχει μία θαυμάσια γενική εικόνα. Είχαμε δραστηριοποιηθεί στις εκλογές, είχαμε στείλει μία αποστολή παρατηρητών, κάναμε πολλές συστάσεις και η δημοκρατική αυτή κοινότητα χρειάζεται τη βοήθειά μας και οικονομικά αλλά και από πλευρά ασφαλείας Οπότε η κατάσταση δεν ήταν ε, η ίδια πριν δύο-τρία χρόνια όταν ο προκάτοχός μου είχε πάει στο Πακιστάν. Δεύτερον, πρέπει να ε, υπάρχει μία προσέγγιση επιβολής ε, του δικαίου διότι στην ΦΑΤΑ στο βορειο, στη βορειοδυτική ε, ε, ε, περιοχή υπάρχουν πολλά προβλήματα η Επιτροπή θα στείλει μία αποστολή για να καθορίσει τι μπορεί να, να συμβάλλει όλο και περισσότερο υπάρχουν προβλήματα για να μπορέσει κάποιος να, ε, να δικαστεί λόγω ελήψεως αποδεικτικών στοιχείων και θα είμαστε πολύ δραστήριοι τέλος όσον αφορά την ε, αστυνομία βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη την πτυχή της δικαιοσύνης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τη την ε, αναπτυξιακή βοήθεια για να βοηθήσουν το Πακιστάν και στην ε, πρόληψη ε, της πιο ριζοσπαστικής αντιμετωπίσεως των θεμάτων και ε, τέλος ένα άλλο πολύ βασικό θέμα που έχει σημασία η κατάσταση στην Αμερική, η ε, εκλογή νέου Προέδρου ο οποίος απεφάσισε να κλείσει το Γκουαντάναμο και να ε, συμβάλλει στην επιβολή του δικαίου θα βοηθήσει στον διατλαντικό διάλογο ότι την περασμένη Δευτέρα οι Υπουργοί είχαν το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και συζήτησαν με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να στηρίξει τους Αμερικανούς να λύσουν το πρόβλημα του Γκουαντάναμου. Αρχικά ήταν ε, μία συζήτηση άτυπη ε, κατά το γεύμα αλλά θέλουμε να διερευνήσουμε και να δώσουμε μία σφαιρική θετική ε, απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως δηλαδή ε, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει αν κάποιος θα γίνει αποδεκτός στο έδαφος ενός κράτους το οποίο είναι κυρίαρχο και πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του αλλά σας υπενθυμίζω το 2002 είχαμε στο Συμβούλιο υιοθετήσει μια κοινή θέση για να ε, ε, να υποδεχθούμε 13 Παλαιστινίους αλλά τότε ήταν ε, παρόλο που ήταν κοινή απόφαση δραστηριοποιήθηκαν 5-6 χώρες μόνο. Τώρα όμως πρόκειται για άτομα τα οποία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι πολύ φυλακισμένοι οι οποίοι πρέπει να επαναπατριστούν στις χώρες τους, θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα αποκαταστάσεως και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να εξεταστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα προωθήσουμε. Τέλος, στο Συμβούλιο ε, Ασφαλείας θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις ε, αρχές ε, τις αρχές προστασίας ιδίως από εκρηκτικά όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Είπατε ούτως ή άλλως ότι θα καλέσετε τον συνάδελφό μου Τζανέλα. Εγώ θα πάω απόψε και αύριο σε ένα σεμινάριο στην Πράγα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα πρώτα στοιχεία ενός πολιτικού πακέτου το οποίο θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο για να καλύψει τρία από τα τέσσερα, τις τέσσερις αρχές για να δούμε πώς θα μπορέσουμε ε, να, ε, να τη, το CPN. Πρέπει να ε, πρέπει να προωθήσουμε τις αρχές ασφαλείας. Η κατάρτιση του προγράμματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μία έκθεση. Και τέλος προσπαθώ να διερευνήσω τι παραπάνω μπορεί να γίνει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ε, χρειάζεται ε, ε, μια επιχείρηση ε, στην EDA ε και θα πρέπει να δώσουμε τις έμπειρες γνώμες μας και να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας και η παρακολούθηση διαθαλάσσης είναι επίσης ένα θέμα που μας ε, απασχολεί και αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα σας παρουσιάσω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή σα. Έχω πρώτος μια ερώτηση. Το θέμα των στρατοπέδων τρομοκρατίας, εκπαίδευσης δηλαδή ε, τρομοκρατών. Η ερώτησή μου είναι πόσοι υπάρχουν εκεί, πόσοι εκπαιδεύονται και τι γίνεται όταν επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Η νομική κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη τι προβλέπει. Εάν κάποιο κράτος, ε, συμμετα... Ε, κάποιο κράτος θεωρεί ότι και η μόνη συμμετοχή σε ένα τέτοιο στρατόπεδο εκπαίδευσης είναι ένα ε, έγκλημα παράπτωμα ή οτιδήποτε. Και ο κ. Μητρακόπουλος έχει μια ερώτηση επίσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κ. Ντεκέρκχοφερ για την παρουσίασή του. Θα σας πω πολύ επιγραμματικά τις ερωτήσεις μας για να μην μακρηγορήσω. Πρώτον, η συλλογή στοιχείων, πληροφορίας και η σχέση τους με άλλες υπηρεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάποια εμπειρογνωμοσύνη στην αντιμετώπιση των πληροφοριών αυτών για τους τρομοκράτες. Δεύτερον, εγκλήματα στον κυβερνόχωρο, κυβερνόχωρο, συγγνώμη, η εξέλιξή τους και η σχέση τους με την τρομοκρατία. Τρίτον, οι σχέσεις μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος ιδίω στον τομέα που αφορά την αγορά εξοπλισμών. Και τέλος, οι διεθνείς σχέσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων μεταξύ τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να έχουμε ίσως ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. Μάλιστα. Η πρώτη σας ερώτηση είναι μια ερώτηση που Αναρωτήθηκα κι εγώ και την έχω υποβάλει σε πολλούς ε, που πήγαν στο Πακιστάν. Υπάρχει ανησυχία στις υπηρεσίες κατασκοπίας. Δεν έχω στοιχεία αριθμητικά. Αλλά όσο πάει και περισσότεροι άνθρωποι πάνε στο Πακιστάν για εκπαίδευση. σε Ισλαμικά σχολεία ή σε στρατόπεδα αυτά εκπαίδευση τρομοκρατία. Αν θυμάσαστε, το Δεκέμβριο, στις 11 Δεκεμβρίου, έγιναν κάποιες ε, ε, συλλήψεις στο Βέλγιο με ανθρώπους που σχετίζονται με το Πακιστάν. Εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα, ενώ στο παρελθόν πριν από πέντε χρόνια ε, το εμπόριο αυτό γινόταν από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη και στο Πακιστάν ε, σχέσεις με την Μεγάλη Βρετανία. Τώρα δεν ισχύει αυτό έτσι απόλυτα. Ξέρετε ότι έγινε νέος ορισμός πριν από μερικές εβδομάδες για να ορίσουμε καλύτερα το θέμα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι διδασκαλία Λίγα κράτη-μέλη προβλέπουν ειδικά δίωξη του γεγονότος ότι κάποιος πάει στο εξωτερικό σε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης για να εκπαιδευτεί. Και συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται κάτι να γίνει, ιδίω όταν ε, μίλησα με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και υπηρεσίας κατασκοπίας ε, στο Πακιστάν. Εκείνοι ελέγχουν όσο μπορούν και νομίζω ότι είναι πολύ καλοί στον έλεγχο αυτό και μπορούν να συνεργαστούν και καταλαβαίνουμε γιατί μόνο εάν υπάρχει εγκληματική πράξη. Δεν μπορούν να ελέγχουν τον τεράστιο ρυθμό ανθρώπων που μπαίνουν στο Πακιστάν για νόμιμους λόγους και εμείς δεν θα το δεχόμασταν κάτι τέτοιο. Έχοντας λοιπόν έναν ορισμό μέσα στο ποινικό δίκαιο που θα καλύπτει αυτή την περίπτωση, θα βοηθηθούμε πάρα πολύ και θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτό που κάνει η Γερμανία σχετικά. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια, γιατί θα πρέπει να συλλεχθούν αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποδείξεις δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συλλεχθούν πάντα. Έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία Όταν κάποιος πήγε σε μια ξένη χώρα και παρακολούθησε μια τέτοια ε, ε, εκπαιδευτική μονάδα μπορούμε να το πούμε γιατί αν γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο πρέπει να το κλείσουμε. Μετά, η σχέση της συλλογή ε, στοιχείων από κατασκοπικές οργανώσεις και από άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει βέβαια, δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω όμως, δεν είμαι ο σωστός συνομιλητής για κάτι τέτοιο, γιατί η συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν διαβάσετε τη συνθήκη της Λισαβόνας βλέπετε ότι το σημείο αυτό τονίζεται. Και η συνθήκη της Λισαβόνας λέει τα ίδια που λέει και η σημερινή συνθήκη ότι είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για την εσωτερική ασφάλεια. Εσωτερική ασφάλεια. και είναι μόνο υπεύθυνε για την εθνική ασφάλεια, κατασκοπία δηλαδή. Βέβαια είμαι παρόν σε πολλές συνεδριάσεις και ομολογώ ότι ήμουν σε διάφορες συναντήσεις όπου διαφάνει ότι η συνεργασία αυτή είναι αρκετά καλή. Υπέβαλα την ίδια ερώτηση στον ε, Πακιστανό επικεφαλή της ΆΙΣΑΙ και έχουν ένα, ένα, μια υπηρεσία κατασκοπίας πολιτικής κατασκοπίας αν θέλει και όχι και βελτιώνουν βελτιώνουν αυτό που κάνουν. Έχουν μια αρκετά καλή συνεργασία με πολλά κράτη-μέλη. Όχι και τα 27 ίσως, αλλά με πολλά. Το ίδιο ισχύει και με τις ε, σχέσεις με τις υπηρεσίες ε, της ε, Βορειοαφρικής. Εγκλήματα στον κυβερνόχωρο. Κρομοκρατία στον κυβερνόχωρο. Πριν από μερικά χρόνια προβλέψαμε κάποια νομοθεσία για να είναι κάτι τέτοιο να θεωρείται έγκλημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Γαλλική Προεδρία ήταν πολύ εδραστήρια το τελευταίο εξάμεινο και υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα στην Ευρωπόλ που συνδέει όλες τις εθνικές σχετικές πλατφόρμες στα 27 κράτη-μέλη για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν έτσι όλες οι σχετικές πληροφορίες για το έγκλημα στο κυβερνόχωρο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη την κατάσταση αυτή. Από όσο ξέρω βρισκόμαστε στην απαρχή του τρομοκρατίας αυτής. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως του τύπου δηλαδή που είδαμε που εμφανίστηκε στην Εσθονία, όπου το ίντερνετ χρησιμοποιήθηκε σαν όπλο. Θα γίνει ένα σεμινάριο την επόμενη εβδομάδα σε καμιά δεκαετία μέρες δηλαδή και συμφωνώ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανωθεί πολύ καλύτερα στον τομέα αυτό. Τώρα, τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα, ιδίω όσον αφορά τα όπλα. Είναι μια πολύ σχετική ερώτηση και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στη Σαχέλ. Γιατί έχουμε κάποια αδύναμα κράτη, για να μην πούμε τίποτα άλλο, και υπάρχουν και ορισμένες ομάδες, οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους Υπάρχουν μακρές συζητήσεις κατά πόσο είναι τώρα σχετίζονται με την Αλκαίδα ή όχι, κάνουν εμπόριο α, όπλων ή όχι. Αλλά πάντως οπωσδήποτε μία επανάσταση σημαίνει ότι χρειάζονται όπλα οι άνθρωποι αυτοί και κάποιο διακανονισμό, α το πούμε έτσι, θα έχουν με εκείνου οι οποίοι ε, δρούν. Υπάρχει λοιπόν συσχετισμό, υπάρχουν σχέσει. είναι σωστό. Τι είπατε ακόμα, συνεργασία μεταξύ των διεθνών ε, οργανώσεων εκτός μικροφώνου ο κ. Δημητρακόπουλος. Α, μεταξύ των διαφόρων ομάδων, σε διεθνέ επίπεδο, των δημοκρατικών ομάδων δηλαδή. Εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση στον κόσμο για την οποία συζητάμε. Αν πάρουμε το Πακιστάν, είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η εικόνα, γιατί θα πρέπει να διακρίνει κανένας μεταξύ εκείνων που ε, απλώς επαναστατούν, παστούν και μετά υπάρχουν άλλες ομάδες, η ΣΥΑ κατά τον ΣΥΑ, παραδείγματος χάρη, ορισμένοι από τους επαναστάτες παστούν έχουν κάποια σχέση με την Αλκαϊντά και υπάρχει συζήτηση κατά πόσον η Αλκαϊντά εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή οργάνωση στο κέντρο ζήτης ή απλώς ε, έχει υποκαταστήματα σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες, οι Ελιτοί, οι και κλπ. Οι οποίες δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένες με άλλες, αρκετά ανεξάρτητες. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε διαμακρόν αυτό. Αλλά δείτε ότι η κύρια απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την Αλκέντα το πυρήνα της ΚΑΙΔΑ ε, όπως είπαμε. Και είναι διαφορετική κατά κάποιο τρόπο από την Αλκαΐδα στο Ισλαμικό Μαγκρέπ. Εγώ δεν βλέπω όμως συγκεκριμένε συνδέσεις μεταξύ του δικτύου αυτού και άλλων οργανώσεων που δρούν στην Ευρώπη, όπως το ΠΚΚ παραδείγματος χάρη, που είναι στο καταλογό μας μια ενεργή οργάνωση, συλλέγει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύντομα θα υποβάλω στο Συμβούλιο κάποιες προτάσεις ε, προς την κατεύθυνση αυτή για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ΠΚΚ στην, στην Ευρώπη γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο ε, συλλέγουν χρήματα για να μπορέσουν να οργανώσουν επιθέσεις ε, στην Τουρκία και στο Ιράκ, αλλά δεν βλέπουν να υπάρχει κανένα συσχετισμό μεταξύ της ΠΚΚ και της Αλκαΐντα, ας πούμε. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προτείνω ε, τώρα να ακούσουμε τους δύο άλλους ομιλητές και ε, να γίνουν οι ερωτήσεις και προς τους τρεις. Ε, μέχρι τις 10 και μισή έχουμε χρόνο, οπότε δεν χρειάζεται να περιοριστούμε και δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Ρόιλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι ήθελα κατερχήν να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή για την Άμυνα και την Ασφάλεια που κάλεσε για πρώτη φορά την Ιντερπόλ σε μια από τις συνεδριάσεις της. Εγώ ως ειδικό εκπρόσωπος, μόνιμος αντιπρόσωπος μάλλον εδώ και έξι μήνες στις Βρυξέλλες, θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό για να εξηγήσω τι έχουμε ως στόχο για το μέλλον. Ο Γενικός Γραμματέας της Ιντερπολ πρόσφατα επισκέφθηκε μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Βομβάης το Πακιστάν και την Ινδία για να εξετάσει τη δυνατότητα ε, αστυνομική συνεργασίας έχουμε. Και επανήλθε με την πλήρη διαθεσιμότητα των τοπικών αρχών να συνεργαστούν ε, με την ε, διεθνή κοινότητα. Όπως επίσης ε, και με τη βούληση των στρατιωτικών να συνεργαστούν. Αν θέλουμε εμείς διεθνή συνεργασία, αστυνομική συνεργασία, πρέπει καταρχήν να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες μας και να διαδώσουμε αυτήν την, να την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό συμβαίνει σε ένα βαθμό και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας είναι να ενισχύσουμε την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε λοιπόν τα δύο. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Θεοφιλόπουλο που ήρθε από τη Λιόν και είναι ένας από τους εμπειρογνώμονές μας για θέματα τρομοκρατίας και να σας αναφέρει ποια είναι τα μέσα και δυνατότητες της Ιντερπολ να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι Βασίλης Θεοφιλόπουλος και είμαι ένα μέλος ε, της υποδιεύθυνσης δημόσιας ασφαλείας και τρομοκρατίας της Ίντερπολ ε, ε, αρκετά χρόνια και επιπλέον ε, είμαι υπεύθυνος για μία task force στο πρόγραμμα Nexus και στην παρουσίασή μου θα παρουσιάσω την θετική και προληπτική προσέγγιση της Ιντερπολ η οποία συγκεντρώνει τις δυνάμεις της ενάντια της τρομοκρατίας ε, στην ε, συγκέντρωση πληροφοριών και επεξεργασία πληροφοριών. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να παρουσιάσω τους στόχους και να τονίσω τα βασικά θέματά μας διότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ε, ε, του καταστατικού της Ιντερπολ προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τις τους τρομοκράτες να τους, προ... καταπολεμήσουμε παντού και να ε, συμβάλλουμε αποτελεσματικά εις ε, την πρόληψη του εγκυρήματος. Η Ιντερπολ έχει παρουσιάσει διάφορα θέματα τα οποία μόνο αυτή μπορεί να παρουσιάσει και ε, προσπαθούμε να ε, στείλουμε στην αστυνομία όσο δυνατόν πιο γρήγορα τις πληροφορίες, να έχουμε ε, διάφορες υπηρεσίες ε, για την εξυπηρέτηση της αστυνομίας και να αναπτύσσουμε τα στοιχεία και είναι πολύ βασικό για όλα τα χρόνια για όλα τα κράτη να ξέρουν ότι στο καταστατικό μας ε, καθορίζεται ότι η Ίντερπολ δεν επεμβαίνει σε θέματα πολιτικά, ε, στρατιωτικά, φιλετικά ή θρησκευτικά. Ε, προσπαθούμε να ε, συνεργαστούμε ακόμη και αν δεν υπάρχουν ε, διπλωματικές σχέσεις μεταξύ κρατών. Στηρίζουμε τα κράτη-μέλη μέσω ενός δικτύου γραφείων. Έχουμε, ένα, έχουμε πέντε γραφεία και ένα γραφείο σύνδεσμος στην Μπαγκόγκο και ένα γραφείο στις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή του 2009 ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του νέου δικτύου μας ε, επικοινωνιών και το οποίο συνδέει τις 187 χώρες μέλη της Interpol. Στο παρελθόν ποτέ δεν είχαμε μπορέσει να συνδέσουμε τόσες πολλές χώρες και να δώσουμε αυτό το εργαλείο επικοινωνίες για την επεξεργασία των στοιχείων. Η κατάρτιση του νέου δικτύου και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών είναι αποτελεσματικές, παγκόσμιες και ασφαλείς και έτσι η Interpol μπορεί να προωθήσει την πρόσβαση σε όλα τα σύνορα, σε όλα τα αεροδρόμια ώστε να μπορεί να έχουμε να πάσα στιγμή επεμβάσεις. Ε, έχουμε ε, ένα πολύ υψηλό αριθμό επεμβάσεων το 2008 ε, και ε, έχουμε μπορέσει να συλλάβουμε πολλούς εγκληματίες τους οποίους ε, είχαμε στην βάση δεδομένων έχουμε ξεπεράσει τις 5.000 συλλήψεις το 2008. Η, η, ε, μέθοδος αυτή παρουσιάστηκε ε, το 2002 για πρώτη φορά και έχουμε ε, περιλάβει στη βάση δεδομένων και ναυτικά φυλάδια και διαβατήρια και ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα τη βάση αυτή δεδομένων εξού και πέρυσι ξεπεράσαμε τα 5 εκατομμύρια α, έρευνες και το 2008 πέραν, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε και περισσότερο. Όλο και περισσότερο μπορούμε να έχουμε επιτυχίες το 2006 πέραν των 2.500, το 2007 πέραν των 6.000 και ε, το 2008 πέραν των 5.000 ε, οπότε κατόπιν ετήσεως των κρατών μελών η Ιντερπόλο μπορεί να ε, ενημερώσει για τους υπόπτους τρομοκράτες ή εγκληματίες έχουμε διάφορα είδη κοινοποιήσεων με διαφορετικά χρώματα και έχουμε και ένα ειδικό έγγραφο το οποίο όμως θα συζητήσουμε αργότερα σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Όσον αφορά ε, την Γενική Διεύθυνση θα ήθελα τώρα εδώ να αναφερθώ ουσιαστικά μόνο στην τρομοκρατία και βλέπετε από το χάρτη αυτή πώς καταρτίζεται ε, αυτή η διεύθυνση. Ε, έχουμε διάφορα τμήματα δημοσίας, ασφαλείας και τρομοκρατίας, ε, καταπολέμησης της διαφθοράς και υπάρχουν και υποδιαιρέσεις στις διευθύνσεις στην, στην υποδιεύθυνση τρομοκρατίας περιλαμβάνονται διάφοροι ε, τομείς ευθυνών για τον βιολογική τρομοκρατία, για το περιβαλλοντολογικό έγκλημα και ούτω καθεξής. Ε, το Σεπτέμβριο 2002 δημιουργήσαμε ε, μία task force για να μπορέσουμε ε, να βοηθήσουμε την Interpol ή στις έρευνές της και έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα περιφερειακά το πρόγραμμα Nexus, το πρόγραμμα Μέσης Ανατορής, το πρόγραμμα Baobab για την Αφρική, το Amazon για την Κεντρική και Νότια Αμερική, ε, ειρηνικός για την περιοχή του Ιρνικού και Ανατολική Ασία και ε, τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σε θέματα τρομοκρατίας. Η πρώτη στόχη αυτής ε, της Task Force είναι να μπορέσει ε, να συγκεντρώσει πληροφορίες κατά τρόπον ώστε να προσφέρει αναλυτικές εκθέσεις προς τα κράτη-μέλη και να ε, τα συνδράμει για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και ε, να έχει ε, και εξομοιατικούς επαφών στα διάφορα κράτη. Στο δίκτυο αυτό προσπαθούμε ε, να παρακολουθούμε όλα τα θέματα που άπτονται της τρομοκρατίας κατά τρόπον ώστε να αντιδρούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά να μπορούμε άμεσα να αντιδρούμε στα μηνύματα και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε μία καλή σχέση ε, και να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μας. Η μονάδα αυτή ε, δραστηριοποιείται σε ε, ε, πέραν των 140 χωρών και βλέπετε ότι το 2008 περιλαμβάνει 201 μέλη δηλαδή βελτιώσαμε το δίκτυό μας και χρησιμοποιούμε επίσης και την ε, ιστοσελίδα μας ε, η οποία περιλαμβάνει και φωτογραφίες και στοιχεία για τους ε, εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω ενός password έχουμε ε, την έδρα στην Νέα Υόρκη για να υπάρχει στενή συνεργασία με ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας και ε, υπάρχει ε, μία ειδική, ε, ένα ειδικό μήνυμα το οποίο εξέδωσε τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την τρομοκρατία και την Αλκάιντα. Έχουμε επίσης πάρα πολλές ενημερώσεις σχετικά με τρομοκράτες οι οποίες δημοσιεύτηκαν το 2008 και έχουμε μία βάση δεδομένων για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προβούν σε έρευνες δίδοντάς τους τις αναγκαίες πληροφορίες, ε, τα στοιχεία των ατόμων και εφιστώντας την προσωπή ε, σε άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε ορισμένες ε, χώρες. Έχουμε στοιχεία σχετικά με το DNA, τα κλεμμένα αυτοκίνητα, τα κλεμμένα διαβατήρια και ούτω καθεξής έχουμε μπορέσει να πολλαπλασιάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο ε, επί 5 από το 2001 τα στοιχεία που έχουμε στη βάση δεδομένων μας. Βλέπετε εδώ πόσα άτομα, ε, πόσοι ύποπτοι είναι καταγεγραμμένοι το 2008 και θα σας δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ε, χωρίς πολλές λεπτομέρειες γιατί συνεχίζεται η έρευνα αλλά πρόκειται για μία έρευνα των Ιταλικών αρχών για διεθνείς διασυνδέσεις είχαμε ε, επιβεβαιωμένες 18 συλλήψεις και ε, οι αρχές του Μιλάνου είχαν εκδώσει εντάλματα συλλήψεως για 20 άτομα εκ των οποίων μπορέσαμε να βρούμε τα 9 μέσω της βάσης δεδομένων μας. Είδαμε ότι ορισμένα από τα άτομα αυτά ήταν, ε, ε, περιλαμβανόντουσαν σε ε, σημειώματα της Interpol και ανακοινώσεις και μπορέσαμε μέσω αυτών να δώσουμε στα κράτη-μέλη επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορούσε τις φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα και να συμβάλλουμε σε πολλές συλλήψεις στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε στη συνέχεια αναπτύξει διάφορα θέματα με την βοήθεια ε, των στοιχείων μας μετά από εθνικές καταστηφές ή μεγάλα διεθνή γεγονότα ε, και έχουμε αναπτύξει και διάφορες ομάδες οι οποίες μπορούν να παρέμβουν αμέσως σε χώρες οι οποίες έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις Χρειάζεται όμως να υπάρξει μία αίτηση και μία ε, άδεια για την χώρα η οποία ενδιαφέρεται και αυτό προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια και επίσης η IRD δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις εθνικές αρχές, απλώς να τις συνδράμει σχετικά με το ο πρόγραμμά μας βιοτύπων η Interpol ε, ε, έχει το πρόγραμμα της βιολογικής τρομοκρατίας και προλήψεώς της και ε, το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει ε, ε, επισήμως το 2005 μέσω ενός συνεδρίου για, για τη βιολογική τρομοκρατία συμμετείχαν στο συνέδριο αυτό 155 χρόνια, χώρες μέσω των ειδικών απεσταλμένων και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Προσπαθήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να ε, τονίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος βιολογικής τρομοκρατίας και δεύτερον να προσφέρουμε εκπαίδευση για ανταπόκριση στην ε, απειλή αυτή. Έχουμε οργανώσει διάφορα εργατιστήρια και ε, ε, περιόδους ε, εκπαιδεύσεως ε, και ε, πρόκειται το, η επόμενη αυτή, το επόμενο σεμινάριο να γίνει 16 με 19 Μαρτίου ή στην Κεντρική Αμερική. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ε, τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε άτομα τα οποία από κοινού μπορούν να εντοπίσουν τις ελλείψεις, να βελτιώσουν την επικοινωνία και ε, να ε, συστήσουν λύσεις για να καλυφθούν τα υπάρχοντα θεσμικά κενά. Έχουμε οργανώσει και δύο ασκήσεις υψηλού επίπεδου αφενός ε, για το πώς μπορεί κανείς να εντοπίσει ε, την απειλή ε, μια τρομοκρατικής ενέργειας και την αντίδραση και δεύτερον να αξιολογήσουμε τις εθνικές δυνατότητες για να προλάβουν την βιολογική τρομοκρατία ε, με τους πόρους και την εφαρμογή των αναγκαίων μεθόδων. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους εθνικούς ε, επικεφαλείς των προγραμμάτων για να συνεργαστούν. Έχουμε τρία μέλη στα προγράμματα για να μπορούν ε, καταρχήν να εντοπίσουν τα όπλα, δεύτερον ε, να παρακολουθήσουν τα ίχνη τους και το τρίτο είναι ε, βαλιστικές πληροφορίες μέσω του δικτύου της Interpol το 2008 έχουμε καταρτήσει έναν πίνακα αναφοράς και η μορφή αυτή επιτρέπει εις τους ερευνητές να εντοπίσουν ένα ε, ε, ένα ε, όπλο προτού ξεκινήσουν την αναζήτηση και δίδουν στον ε, ερευνητή ε, συγκεκριμένα στοιχεία καθώς επίσης ε, και ένα πολύ ψηλό αριθμό εικόνων υψηλής ποιότητος διατίθενται δε γαλλικά και αγγλικά. Αυτή η αίτηση πληροφοριών για τα όπλα επιτρέπει εις ε, τις ε, αρχές να έχουν το ιστορικό αυτών των όπλων ε, το δίκτυο το οποίο έχει καταρτιστεί ε, επιτρέπει να εντοπίσουμε τα βαλιστικά αποτυπώματα τα οποία αφήνει κάθε όπλο και η τεχνολογία μας επιτρέπει να συγκρίνουμε χιλιάδες τέτοια αποτυπώματα εντός ορών αλλά δεν υπάρχει ακόμη ένα δίκτυο για την διεθνή σύγκριση ε, και ε, παράθεση των στοιχείων έχουμε 45 χώρες οι οποίες έχουν τη σχετική τεχνολογία και συνεργάζονται με την Interpol και ελπίζουμε ότι η ανάλυση αυτών των βαλιστικών στοιχείων θα μπορέσει να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε τις διαδρομές που ακολουθούν τα όπλα και οι λαθρέμποροι. Ε, επ' αυτού υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία όλων των δεδομένων μας όπως σας είπα είναι το άρθρο 2 και 3 του καταστατικού της Ίντερπολ και οι πληροφορίες, ε, η προστασία πληροφοριών για την αστυνομική συνεργασία και ε, υπάρχει ένα νομικό νομική υπηρεσία της Γενικής ε, ε, της ε, Γενικής Γραμματείας και μια δεύτερη υπηρεσία. Νομίζω ότι αυτή ήταν η παρουσίασή μου και είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε δεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην υποβολή ερωτήσεων. Ο πρώτος θα είναι ο κύριος Βιαλοβιέσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευγνωμονώ ιδιαίτερα κύριε συντονιστά και κύριε εκπρόσωπε της Ιντερπολ για τις ε, τόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με δράσεις που ελπίζω ότι θα είναι αποτελεσματικές. Έχω δύο ερωτήσεις. Ο συντονιστής μας είπε ότι στην Ισπανία προσπαθούν να μετριάσουν την, ε, τον παλμό των ε, ε ημάμιδων ε, ε στις στις διάφορες σχολές ή τζαμιά. Εγώ γνωρίζω πολλούς μουσουλμάνους γερωμένους και στη Γαλλία και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Είπατε ότι γίνονται και προσπάθειες στην Ινδονησία, στο Μαγκρέμπ, στο Μαρόκο. Αλλά να ρωτήσω. Σαουδική Αραβία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τους στο Αφγανιστάν, στους ε, Παστούν, αλλά και στο Πακιστάν και στη Μαλαισία και στην Ινδονησία στις Ισλαμικές σχολές οι Ουαχαβίτες ε, δάσκαλοι από τη Σαουδική Αραβία είναι αυτοί που είναι φημισμένοι και είναι και καλοί διαδάσκαλοι. Βέβαια δεν είναι τρομοκράτες, αλλά ε, είναι ένα ιδεολογική πίεση ασκούνε διότι διδάσκουν το πιο σκληρό, το πιο αδιάλακτο Ισλάμ και οι νέοι που αποφυτούν από αυτές τις Ισλαμικές σχολές μετά στρατολογούνται από την Αλκάιντα. Γίνεται κάτι μέσω του Αραβικού Συνδέσμου ή τέλος πάντων κατευθείαν με τη Σαουδική Αραβία που είναι και ελαφρώς σύμμαχος με τη Δύση γίνεται κάτι. Μπορούμε να ε, περιορίσουμε αυτή την επιρροή των ουαχαβητών στην ε, νεολαία πολλών χωρών. Τώρα πριν από τρία χρόνια ως ε, που συμμετείχα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, συμμετείχα στη Λισαβόνα σε μία συνάντηση για το οργανωμένο έγκλημα και ήταν πολύ απεσιόδοξη αυτή η συνάντηση διότι οι εκπρόσωποι της αστυνομίας, των δικαστών, των εισαγγελέων κτλ. απέδειξαν πριν από τρία χρόνια σας λέω, απέδειξαν ότι εμείς ε, είχαμε χάσει το τρένο ότι το οργανωμένο έγκλημα ε, είχε προχωρήσει πολύ. Είχαμε, έχουμε τεχνολογικές πρόοδους, ε, νέες οργανώσεις που εμφανίζονται. Εγώ λοιπόν προτείνω συγκρίνοντας και με το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν είναι απλά και μόνο μία χώρα, είναι μία μεγάλη ήπειρος. Προτείνω να έχουμε αυτήν τη συνεργασία της αστυνομίας βασιζόμενη στην κοινή νομολογία και στη Λισαβόνα αποδείξαμε ότι ήμασταν πάρα πολύ καθυστερημένοι κυρίως έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν κύριε σύντονιστα τι κάνουμε, προχωράμε πέρα δηλαδή από τους αστυνομικούς ε, και τους ε, δικαστές και από τις χώρες οι οποίες δεν ήθελαν έγκαιρα να ανακοινώνουν τις πληροφορίες τους. Τι λέτε, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Ευχαριστώ. Δυστυχώς έχουμε περιορισμένο χρόνο. Παρακαλώ να περιορίσετε τις τοποθετήσεις σας στα δύο λεπτά. Ο κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχει άμεση σχέση με την ε, τωρινή ε, συνάντηση. Θα ήθελα όμως να συγχαρώ τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε αυτή η υποεπιτροπή να καταστεί επιτροπή με πλήρης αρμοδιότητες στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία διότι η διάσταση του, του, θέματος είναι, τεράστια διότι επίσης ε, εμάς ε, μας στοιχίζει ιδιαίτερα ως βουλευτές ε, το να χρειάζεται να κάνουμε τη διάκριση ποια από τις συνεδριάσεις θα πάμε, διότι συνεδριάζει ταυτόχρονα με άλλες επιτροπές. Κύριε συντονιστά, άλλαξε μια κατάσταση πολιτικά πάρα πολύ σημαντική και μιλάω για τις αλλαγές στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου και η κυβέρνηση άλλαξε αλλά και η πολιτική ε, η αντιτρομοκρατική πολιτική. Δεν λέω ότι μειώθηκε η σημασία της τρομοκρατίας, είναι η ίδια που είναι και για μας. Αλλά τέλος πάντων σταμάτησε αυτή η διάχυτη ιδεολογία του απόλυτου κακού κτλ. Και η Προεδρία Ομπάμα μιλάει περισσότερο για πρόληψη, για διάλογο. Πέρα από τα μέσα intelligence και συντονισμού με την Ευρώπη. Πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη με αυτή τη νέα κατάσταση. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουμε ακριβώς το άκρο αντίθετο Δηλαδή ας πούμε, αντιμετωπίζεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μόνο μέσα από το πρίσμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει όμως να είμαστε και αποτελεσματικοί, δηλαδή συντονισμός αστυνομίας, των δικαστών, αποτελεσματικότητα στη σύλληψη και καταδίκη των τρομοκρατών. Επίσης ε, και το θέμα του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών που ξεκίνησαν η Τουρκία με την Ισπανία μέσα από τη συμμαχία των πολιτισμών που αποτελεί πλέον ε, κομμάτι των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα πλέον δηλαδή ε, κομμάτι για ε, που εντάσσεται στη λογική της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και εργαζόμαστε στο, στην πρόληψη του μέλλοντος της τρομοκρατίας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Συνάδελφος έχει το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τεκερχόπ. Δύο πράγματα. Πρώτο, Αναφέρεται για την ανάπτυξη τρομοκρατικών ε, δραστηριοτήτων στην περιοχή του Σαχέλ ε, που ίσως είναι και ανακατεμένη η Αλκάιδα αλλά δεν είναι μόνο το, ε, το Σαχέλ αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι της Σαχάρας στην Αλγερία Λοιπόν, εσείς τι λέτε, ε, ε, ε, μέσω οι δορυφορικές σας φωτογραφίες επιβεβαιώνουν τέτοια πράγματα. Επίσης είπατε, πριν από την Γάζα είχε υποβαθμιστεί η εικόνα των φανατικών Ισλαμιστών. Τι λέτε όμως εσείς σήμερα. για την αντίδραση της κοινή γνώμης υπέρ του ΑΜΑΣ και το πώς ε, το βλέπουν αυτό οι αραβικές χώρες και τι θεωρείτε ότι άλλαξε στην τρομοκρατία συνολικά. Κύριε Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντεκερκόβε. Ξέρω ότι στην δήλωσή σας είπατε ότι ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να ασχοληθούν με τις επιπτώσεις ασφαλείας ε, εάν ε, υποδεχθούν ε, τους κρατουμένους του Κουαντάναμο τους οποίους θα ελευθερώσει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις. Είναι δυνατόν να αντεπεξέλθουμε ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί ως αθώοι από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά έχουν κατά τη συνέχεια ε, υποστεί ε, βασανισμούς και τα λοιπά. Επίσης ε, όσον αφορά το ε, ε, ε, τους Παλαισινίους και την, την Εκκλησία της Γεννήσεως και τα προβλήματα το 2003. Τι πιστεύετε σχετικά με τους κινδύνους για το Σαχέλ και τη Σαχάρα. Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει μία συνεχής διαμάχη στο, στη Σαχάρα και νέοι οι οποίοι μπορούν να εξοπλίσουν ε, ε, την τρομοκρατία, τι, πιστεύετε. Επίσης μπορείτε να μας πείτε πώς θα μπορέσετε ε, να, υπάρξει, να βοηθήσετε στο να υπάρξει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Αυτό θα μπορέσει επίσης να συμβάλλει ε, εις το να ακυρώσουν όλα τα κράτη-μέλη την, ε, ε, την συνθήκη κατά της τρομοκρατίας. Και τελευταία ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας η Europol τι χρειάζεται για να γίνει πιο αποτελεσματική και να συνεργαστεί με την Ιντερνετ Ιντερπόλ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. πάμε στον συνάδελφο Κόνερτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να στραφώ με τις ερωτήσεις μου και τις παρατηρήσεις μου στον κύριο Δεκέρκοφ. Καταρχήν μια συμπληρωματική ερώτηση βάσει αυτό που ακούσαμε εδώ, αναρωτιόμαστε πόσο έντονη είναι η συνεργασία με τη Ρωσία. Τις τελευταίες μέρες η ρωσική πλευρά αναφερθήκε πάλι στην ε, σημασία της, ε, ε, της συμβολής της Δύσης στο Αφγανιστάν και η συνεργασία με το Κάφκασο προτείνανε και διάφορα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αυτή η συνεργασία πόσο λειτουργεί. Δεύτερον, η αντιμετώπιση των τρομοκρατικών ομάδων. Νομίζω το θέμα είναι πάρα πολύ επί, ε, ε, επίκαιρο αυτή τη στιγμή γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να κλείσει το στρατόπεδο του Γκουαντάναμο. Το χαιρετίζουμε αυτό φυσικά, αλλά θα ήθελα, επειδή αναφερθήκατε σε θέματα παιδικού δικαίου, να τονίσω ότι πράγματι πιστεύω ότι ε, όταν κλείσει αυτό το, το στρατόπεδο αρχίζουν μάλλον τα ερωτηματικά να παρουσιάζονται. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν. Τι θα γίνει με την περιθώρια εξέλιξη παραδείγματος χάρη του ποινικού δικαίου. Κατά πόσον από της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής υπάρχει θέμα ποινικού δικαίου αν κάποιος εκπαιδεύεται τρομοκράτης. Πόσο υπάρχει κάτι τέτοιο, πόσο μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε. Αναφερθήκατε σε κάποιες πρώτες κινήσεις του Συμβουλίου, αλλά εμείς αναρμοζόμαστε τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ποια θα είναι η νομική βάση για να μπορέσετε εσείς να δράσετε όπως το θέλετε, ούτως ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα αστυνομικά μέτρα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της εξέλιξης του ποινικού δικαίου είναι επίσης ενδιαφέρον εάν ε, σκεφτούμε ότι θα πρέπει να ε, εξελιχθεί και το δίκαιο πολέμου γιατί εδώ έχουμε να αναρτηθούμε πρόκειται για στρατιώτες με τους οποίους έχουμε να κάνουμε, πρόκειται για ένοπλους, ε, ένοπλους ε, πολίτες οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκληματίες ή ακριβώς τι γίνεται. Αν δεν μπορούσαμε νομικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή σωστά, δεν θα μπορούν να είναι αποτελεσματικά καθόλου τα αστυνομικά μέτρα. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξάσουμε το θέμα του ποινικού δικαίου και της ε, εξέλιξής του. Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν αναφέρεστε σε αυτό το θέμα της περιτορυξίας του δικαίου. Ευχαριστώ. Ο συνόλυβος Ρόφσινγκ έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εντυπωσιάστηκα από το δίκτυο που μας παρουσιάσετε σαν δίκτυο ασφαλείας. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον αυτό το δίκτυο ασφαλείας έχει ε, υποστεί εισβολές στο παρελθόν και τι γίνεται με τις πληροφορίες που συλλέγονται. Κατά πόσον υπήρξαν οι εισβολές στο δίκτυο αυτό, κάποιοι που δεν είχαν την άδεια να μπουν στο δίκτυο μπήκανε, έγινε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση, την κατανοήσατε? Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Πολλοί έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στο δίκτυο αυτό. Μήπως κάποιοι καταχράστηκαν τις πληροφορίες ή δόθηκαν πληροφορίες σχόλια να υπάρχει άδεια να χορηγηθούν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Η Βαρόνι Λάτφαντ πολυ η λατφα λατφαντ εχει το λόγο. Τα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε γιατί δεν ήμουν παρούσα να ακούσω την παρουσίαση του κ. Κέρκοφ, γιατί ήμουν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση όσον αφορά το ποινικό δίκαιο επίσης, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε μια κατάσταση στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ιδίως η νομικοί συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών, ήρθαν στις Βρυξέλλες και προσπάθησαν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζω χωρίς επιτυχία, ότι χρειάζεται να ακολουθεί κάποιος τρίτος δρόμος για να μην περνάνε απαραίτητος από τους συνήθεις οδούς του ποινικού δίκαιου όσον αφορά το συσχετισμό των ε, ε, διώξεων ε, ποινικών ε, διώξεων θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την ποιητική δίωξη των τρομοκρατών. Υπάρχει προοπτική αυτή η συζήτηση να μην γίνεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ατλαντικά, όσον αφορά ποιε είναι οι προκλήσει, όσον αφορά αυτή την συνήθη δίωξη σε συνήθη δικαστήρια των υπόπτων τρομοκρατών. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε 50 επιτυχείς δίκες και καταδίκες των δημοκρατών, ανθρώπων που φυλακίστηκαν. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αν υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις, πώς μπορούμε να προσπαθούμε ούτως ώστε να έχουμε τα συνήθεια δικαστήρια να εμπλακούν στην δίωξη αυτών των, των γνωρίζοντας βέβαια το πόσο ευαίσθητα είναι κάποια αποδεικτικά στοιχεία, οι πηγές κλπ, θα πρέπει να βρεθούν κάποιες ένομες λύσεις για αυτή την κατάσταση. Για να μην ακολουθήσουμε την άγουσα αυτή που μας οδηγεί σε ειδικά δικαστήρια, ε, στρατιωτικές επιτροπές, ε, προληπτική σύλληψη. Δηλαδή ή θα πρέπει να δικαστούν οι άνθρωποι αυτοί ή θα πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις ΗΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει αυτός ο διάλογος και να μην έχουμε τον παλιό διάλογο που θα ξεπεράσουμε και θα ανοίξουμε παραθυράκια στην ένωμη τάξη. Ευχαριστώ. Κύριος Δακιαρκόπα, σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρώτη ερώτηση του κ. Βεροσκή όσον αφορά το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας αφενός και αφετέρου μια γενική, γενική απάντηση για το πώς αντιμετωπίζουμε το οργανωμένο έγκλημα. Καταρχήν, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Γιατί βέβαια ε, δεν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει σύνθεση μεταξύ θρησκείας και τρομοκρατίας. Είχαμε μια συζήτηση ε, πρόσφατα όσον αφορά ε, την πιο ριζοσπαστική αν θέλετε κίνηση που υπάρχει εδώ και εγώ χάρηκα που υπήρχε μια συνένεση. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Κατά βάση όμως υπάρχει μια συνένεση όπου το Ισλάμ χρησιμοποιείται πραγματικά για ιδεολογικούς και εγκληματικούς λόγους και δεν σχετίζεται όλο αυτό καθόλου με την θρησκεία αυτή καθ' Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Το ότι υπάρχει κάποια ριζοσπαστική ερμηνεία του Ισλάμ, άσχετα από την τροκοματία όμως, είναι αληθές. Και είναι σημαντικό και εδώ να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια συζήτηση. Ό,τι μπορεί να συμβάλλει σε έναν ε, διάλογο μεταξύ των θρησκειών ότι μπορεί να συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση και σε μετριοπαθή προσέγγιση κατά γνώμη μας είναι θαυμάσιο. Κάποιο νομίζω εδώ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της Ισπανίας και του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, ε, τη Συμμαχία των Πολιτισμών. Εγώ πιστεύω σε κάτι τέτοιο πάρα πολύ Έχω κινητοποιηθεί μάλιστα για να υπάρχει μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Χαβιέ Σολάνα και της ε, Μπενίτα Φεραβανέρα από την άλλη μεριά για να ενδυναμωθεί πραγματική αυτή η συνεργασία, αυτή η συμμαχία στο, ευρωπαϊκό εσωτερικό της Ένωσης. Παραδείγματο χάρη, σκέφτομαι την εργασία που γίνεται για να επιτρεπεί μια ειρηνική αντίδραση εάν υπάρχει, αν μπορώ να το πω έτσι, αύξηση θερμοκρασίας μετά από κάποια ε, ταινία που ε, προκαλεί το Ισλάμ όπως ε, εκείνη η Ολλανδική ταινία ή αν υπάρχει πάλι μια, ένα πρόβλημα με γελιογραφίες όπως είχαμε στην περίπτωση της Δανίας κλπ. Λοιπόν, εμείς υποστηρίζουμε τη συμμετοχή αυτή. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω οποιαδήποτε μορφή διαλόγου, ιδίως με την Σουηδική Αραβία, που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει όπως το είπατε Χθε είχα την ευκαιρία να συναντήσω 25 πρέσβες της Σαουδικής Αραβίας από όλη την Ευρώπη που είχαν έρθει εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σας. Ε, είναι λιγάκι τώρα το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνης. Τα 13 τελευταία χρόνια συμμετείχα στην προετοιμασία των περισσότερων πολιτικών της ε, εσωτερικής πολιτικής, ε, πολιτικής ασφαλείας και πραγματικά θαυμάζω που σε 15 χρόνια πέρασαμε από μια διακυβερνητική συνεργασία ισχυρή όπου τα κράτη-μέλη όμως δίσταζαν εναντί της, ε, ε της Ένωσης των Βρυξελών, δηλαδή από την ε, θέση ισχύ της ειδίκης του Μαστρίχ του 1993 μέχρι να φτάσουμε να έχουμε ένα ειδικό πυλώνα για την εσωτερική αυτή συνεργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνθήκη τη Ρώμη το 1957 προέβλεπε μια κοινή αγορά. Και ακόμα συζητάμε τώρα την τελειοποίηση τη ιστορικής αγορά. Τώρα, αν το συγκρίνουμε αυτό με 15 χρόνια, να πείσουμε τις, όλες τις χρόνες όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας σε εσωτερικό επίπεδο και επίπεδο ποινική δικαιοσύνη είναι θαυμάσιο αυτό, είναι εντυπωσιακό. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη είναι καταπληκτικό. Δέκα χρόνια χρειάζεται να περάσει ο Ρωσίδαντα από το Λονδο, Λονδίνο συγγνώμη, στο Παρίσι. 42 μέρες όμως μόνο για να περάσει κάποιος από τους τρομοκράτες του Λονδίνου από τη Ρώμη στο Λονδίνο. Καταπληκτική πρόοδος, εντυπωσιακή που οφείλεται στο Γεωροζού στην Ευρωπόλ. Ε, στα 15 αυτά χρόνια φτάσαμε στα όρια αυτό που μπορούμε να κάνουμε ομόφωνα. Δεν μπορούμε πια να εργαστούμε πια ομόφωνα για να προχωρήσουμε στο ποινικό δίκαιο. Χρειαζόμαστε περισσότερο. Ομόφωνα είναι αδύνατο. Και άμα δούμε πραγματικά την φιλοδοξία των ε, κοινών ε, αποφάσεων, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι θαυμάσιο, το, η ευρωπαϊκή απόφαση για τη συλλογή των ε, αποδεκτικών στοιχείων κατευνούμενη αποτυχία. Χρειάζεται λοιπόν, θα έλεγα, συναπόφαση. Κατεπηγόντω στα θέματα αυτά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί στη διαδικασία αυτή. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, η συνθήκη τη Λισαβόνη κατά βάση και πραγματικά με δημοσίευσε η συζήτηση που έγινε στη Γαλλία ε, για το δημοψήφισμα δεν είπαν ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα είναι η ε, ευρωπαϊκή διάθεση του τρίτου πυλώνα. Δεν σας λέω ότι άλλα θέματα δεν ήταν σημαντικά, αλλά αυτό ήταν η μεγαλύτερη καινοτομία θα έλεγε. αυτό είναι πρωτής σημασίας. Σε, μια, σε ένα πλαίσιο ομοφωνίας δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είμαι επιπισμένος γι' αυτό. Ο του κ για τι αλλαγέ στις ΗΠΑ. Πραγματικά πρόκειται για μια ριζοσπαστική αλλαγή και μια αλλαγή που ευχόμαστε όλοι να γίνει. Η κυρία Λούτφορντ αναφέρθηκε σε παλιάς μόδας, old fashion είπε, μέθοδο. Η ευρωπαϊκή μέθοδος είναι αυτή και ήταν παλιότερα επίσης η αμερικανική μέθοδος. Εν τω μεταξύ υπήρχαν όμως πολλά πράγματα σκοτεινά που έγιναν που καταρχήν είναι ασύτικα αλλά από την άλλη μεριά, όλα κατεδεικνύουν ότι αυτό που είχε γίνει μέχρι στιγμής όχι μόνο ήταν κατά των αξιών μας αλλά δεν ήταν και αποτελεσματικό. Δεν ε, προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα έλεγα λοιπόν ότι το γεγονός ότι οι ΙΠΑ επανέρχονται στην παλιά τους μέθοδο, στην παλιά τους τακτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι πολύ καλά συνεργαστήκαμε με τις ΣΥΠΑ τα τελευταία χρόνια. Δεν ε, μας άρεσε αυτό που γινόταν, αλλά κάτι μπορέσαμε να καταφέρουμε και θα εμβαθύνουμε τώρα τη συνεργασία, φαντάζομαι. Και προσωπικά έχω να σας πω ότι εάν η Ευρώπη μπορεί να δώσει συλλογικές απαντήσεις στο κλείσιμο του Γκουαντάναμο θα αρχίσουμε τη συνεργασία αυτή με την ε, κυβέρνηση Ομπάμα με το δεξί πόδι και θα μπορέσουμε έτσι να ε, συμβάλλουμε στον, στο διάλογο. Και θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε η κυρία Λόρφορ, ότι εάν μπορούμε να δώσουμε μια συλλογική και κοινοτική απάντηση, έχουμε ένα στοιχείο σημαντικό σε μια πιο ευρεία συζήτηση, γιατί δεν είναι μόνο το Γκουαντάναμο. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει το Γκουαντάναμο και να πάει σε, ευρωπαϊκό, σε αμερικανικό έδαφος και έχουμε και τα θέματα της ε, υποδομής κλπ. Νομίζω ότι απάντησα στην ερώτηση για το διάλογο των ε, πολιτισμών και στην ε, πρόληψη και στο ερώτημα του κ. Γιάνναση, αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο. Στην ιστορία κανένας δεν μπορέσει ποτέ να καταπολεμήσει την τρομοκρατία πλήρως με αστυνομικά μέτρα. πρέπει η τρομοκρατία να χάσει την υποστήριξή στον πληθυσμό, στους πολίτες. Ε, προς τον κύριο έχω να πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι η εξέλιξη Αλγερία είναι ανησυχητική και όταν δούμε πώς κυκλοφορεί στο Ισλαμικό Μαγκρέβι η Αλκαίδα με μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Κάτι πρέπει να συζητήσουμε εκεί με τις αλγερινές αρχές. Τα μεγάλα ερωτήματα που έχουμε στην προετοιμασία της στρατηγικής αυτής της Σαχέλ είναι ποιο θα είναι το ειδικό πλαίσιο προτιμησιακής συνεργασίας, ξέροντας ότι η, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν η Αφρικανική Συγγνώμη Ένωση δεν συμπεριλαμβάνει το Μαρόκο. Ε, ότι δεν είναι όλες οι χώρες σε όλες οι οργανώσεις, δηλαδή χρειαζόμαστε να φτάσουμε σε κάποιο στάδιο, να συζητήσουμε με τους Αλγερνούς και με τους Λιβύους επίσης, που έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Για τη Γάζα δεν θα ήθελα να απαντήσω. Αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζεται άμεσα από τον προϊστάμενό μου, από τον Χαβιά Σολάνα. Είναι Πράγματι, όταν πήγα στο Ισλαμαμπάτ και το είπα στην Επιτροπή Προσωπικών Ελευθεριών, η Αλτζαζίρα στα αγγλικά είναι μια ε, τηλεόραση που είναι αντικειμενική, αλλά 24 ώρες το 24ωρο μεταδίδει εικόνες που δεν ξέρουμε στην Ευρώπη, δεν βλέπουμε στην Ευρώπη και που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όσον αφορά το θέμα του κοντάνα και τι επιπτώσει στην ασφάλεια, αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να προτείνω ότι δεν υπάρχει κοινοτική θέση. Υπάρχει μια συνένεση για να προχωρήσουμε προς την κοινοτική θέση. Αλλά ό,τι και να γίνει, ε, θα γίνει όταν είμαστε έτοιμοι να το μεταβάσουμε αυτό. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν τρεις κατηγορίες κρατουμένων στον Κοντάναμο. Οι πιο επικίνδυνοι εκείνοι που θα δικαστούν και κατά πάσα πιθανότητα θα καταδικαστούν γιατί υπάρχουν αποτεκτικά στοιχεία για το πόσο επικίνδυνο είναι. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι προληπτικές κρατήσεις όπου δεν ε, έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία γιατί τα αποδεικτικά στοιχεία συλλήφθηκαν μέσω βασανιστήριων κλπ. Οπότε μπορεί να ε, απελευθερωθούν από ένα άλλο δικαστήριο γιατί δεν ήταν σωστά τα στοιχεία αυτά, δεν ήταν σωστός ο τρόπος με τον οποίο συλλέχθηκαν δηλαδή. Μετά, η τρίτη κατηγορία είναι εκείνο που δεν επικίνδυνε, βρέθηκαν ίσως στον ε, άσχημο τόπο σε άσχημη στιγμή. Και για λόγους όμως ε, ε συγκεκριμένους δεν μπορούν να αποστανούν πίσω στις πατρίδες τους γιατί ίσως θα είναι εκεί θύματα βασανισμών και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και θα πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη ε, αποφάσεις μήπως θέλουν να τους υποδεχτούν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται όμως κάποια ε, ασφαλείας. Ίσως κάποια όμως ε, ψυχολογική ενίσχυση αν κάποιος έχει μείνει 7 χρόνια στο Γκαντάναμο, κάποιος διακανοσμό για να είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δεν είναι επικίνδυνοι κλπ. Αλλά αυτά είναι όλα θέματα που οι οι υπηρεσίε κατασκοπία και ασφαλεία ξέρουν πώ θα αντιμετωπίσουν, γιατί υπάρχουν στο παρελθόν και άλλα παραδείγματα. Είναι ακριβό βέβαια, κοστίζει. Για τη Λισαβόνη απάντησα. Για τη Σαχέλ. Ε, το κύριο θέμα που τίθεται εδώ είναι η άμεση επίπτωση της Αλκαίδα του Ισλαμικού Μαγκρέπ στην Ευρώπη. Το ΖΕΙΑ τη δεκαετία του 90 θα θυμόσαστε ότι είχαν υποστηρίξει μια ομάδα στην ε, Γαλλία και ξαφνικά όλοι αυτοί ε, πέρασαν σε άμεση δράση κατά της Γαλλίας. Ξέρουμε ότι η Αλκαίδα υποστηρίζει ορισμένα ε, κυψέλες αν θέλετε στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να περάσουν σε δράσεις άμεσε. Ρωσία. Την ερώτηση του κυρίου Κόνραντ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε συνεχείς επαφές και συναντήσεις με τη Ρωσία. Έχουν εμπειρία στο Αφγανιστάν, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά πάντως πολλά ξέρουν για τη χώρα αυτή και μπορούμε να, τους, ε, να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις τους, ε, να συνεργαστούμε μαζί τους, ε, τι γίνεται με το θέμα των ναρκωτικών, τα διά, οι διάφορες οδοί μέσα στον περνάει η ηρωίνη που έρχεται στην Ευρώπη. Πραγματικά αυτό πρέπει να εξελιχθεί βέβαια και εγώ έχω μια προσωπική σχέση με τον Ρώσο συντονιστή. Έχουμε μια τρόικα την επόμενη εβδομάδα με την Προεδρία, την Κομισιόν και τη Ρωσία. Και όσον αφορά το θέμα της δίδυσης των δικτύων και της διαρροές. Πάνω σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ δεν είμαι στην πρώτη γραμμή δράσης. Για τις διαρροές δεν νομίζω. Για τη δίδυση φοβούμαι ότι ναι. Ε, δεν μπορώ να σας απαντήσω όμως. Το ερώτηση Σαρα Λούτφορτ για την προοπτική μιας ε, διατλαντικής ε, συζήτησης. Εν μέρει απάντησα στην ερώτησή σας. Ένας τρόπος για να έχουμε στενή και φιλική και έντονη σχέση είναι ακριβώς αυτό που είπα και για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο. Αλλά βέβαια υπάρχει ένας διάλογος και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς εκείνοι επιστρέφουν στην παλιά ε, πολιτική. Είναι δύσκολο το θέμα λοιπόν. Τελειώνοντας, ε, σχετικά με το ποινικό δίκαιο γιατί πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτόν αν το ποινικό δίκαιο είναι προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της τρομοκρατίας ή χρειάζεται κάτι παραπάνω είναι ένα δύσκολο ερώτημα την επόμενη εβδομάδα έχω κληθεί στο κοινοβούλιο του Βελγίου για να συζητήσουμε στο θέμα αυτό διότι πολλοί θεωρούν ότι έχουμε υπερβεί τα όρια σχετικά με την τρομοκρατία και μπορεί να διακινδυνεύουν οι προσωπικές ατομικές ελευθερίες και συνδικαλιστικές ε, ελευθερίες. Πρέπει να δούμε όμως εάν το σύστημά μας είναι καλό. Πιστεύω ότι αν υπάρχει μια καλή νομοθεσία η οποία σέβεται τα βασικά ε, ε, τα βασι, τις βασικές ελευθερίες πηγαίνουμε καλά διότι εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπάθησαν να, βγουν εκτός δικαίου ήταν διότι πίστευαν ότι το δίκαιό τους δεν ήταν προσαρμοσμένο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε προσαρμοσμένα μέσα για το δίκαιο και αυτό τίθεται όταν μιλούμε για το εξωτερικό. Δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να φυγεί αμέσως γιατί μόλις έχουμε ε, τελειώσει μια συζήτηση για διεύρυνση και το θέμα της τρομοκρατίας αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μία άσκηση σε πέντε ε, κράτη συγκεντρώνοντα τους βασικότερους νομικούς και δικαστές σχετικά με το θέμα αυτό και σε ένα ενάμιση χρόνο θα παρουσιάσω τα, τις νομικές ελλείψεις διότι πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν σχέση ε, με το χώρο και θα δούμε αν υπάρχουν ελλείψεις αλλά πολύ σωστά λέμε ότι είναι ένα βασικό θέμα διότι διαφορετικά θα υπάρχουν εκτροπές και συγχρόνως θα πρέπει να έχουμε βασίσει την νομοθεσία μας στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ κύριε Ντεκερκό. Τώρα είμαστε σε μια δύσκολη θέση διότι έχουμε και τη συζήτηση με το Συμβούλιο και ε, για, το, για την Ίντερπολ έχουμε ελάχιστο χρόνο για να μας απαντήσετε σε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσω αμέσως ε, ή τουλάχιστον στα θέματα που έθιξε ο κύριος Ντεκερκόβε διότι αυτός ήταν ο κύριος αποδέκτης ερωτήσεων όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που μπορεί να δώσει η Ιντερπολ στην Ευρώπη. Ήθελα να σας πω ότι 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη της Ιντερπολ. Οπότε στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί κατά τη γνώμη μας να ενισχύσουμε την συνεργασία ιδίω όσον αφορά την ε, οδηγία πλαίσιο η οποία αυτή τη στιγμή ε, προχωρά για τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διεθνών οργανώσεων. Αυτό εσωτερικά. Εξωτερικά, εάν μιλάμε για συνεργασία με χώρες σαν τη Ρωσία ή άλλες χώρες ανά τον κόσμο, θα διαπιστώσατε ότι το δίκτυο της Interpol σε 187 χώρες θεωρείται ότι μπορεί να συμπληρώσει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σε σχέση με αυτές τις χώρες. Και δεύτερο μικρό θέμα, εάν κατάλαβα καλά, υπάρχει κάποιος ο οποίος ανέφερε στην εισχώρηση των δικτύων. Δεν ξέρω αν εννοούσε τα δίκτυα ε, της αστυνομίας και συγκεκριμένα τις βάσεις δεδομένων της αστυνομίας είναι, προφανώς ότι, είναι προφανές ότι προστατεύονται και ούτε ένα φυσιολογικό άτομα ούτε εγκληματίες μέχρι στιγμής έχουν διεισδύσει σε αυτά τα δίκτυα. Όσον αφορά την συνεργασία της Interpol και της Europol θα απαντήσει ο κύριος Θεοφιλόπουλος σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Europol και Interpol. Έχουμε στενή συνεργασία ουσιαστικά όμως για την τρομοκρατία σχετικά με το ερώτημά σας. Η Interpol έχει καταρτήσει μία σειρά βάσεων δεδομένων με πολλές πληροφορίες για την τρομοκρατία και περιλαμβάνει στην ε, ε, βάση αυτή δεδομένων όχι μόνο πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και για άλλες ε, χώρες. Οπότε βλέπετε πολλές πληροφορίες που δεν προέρχονται μόνο από την Ευρώπη αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια διεθνής βάση δεδομένων και περιλαμβάνει στοιχεία όχι μόνο για μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά διεθνώς. Ευχαριστώ. Ε, πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ τους πάντες και κλείνει αυτό το σημείο της συζητήσεως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αντιλαμβάνουμε ότι ακόμη ασχολείστε με την τρομοκρατία, αλλά σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε τις συζητήσεις σας και οι συζητήσεις αυτές να συνεχίσουν ενδεχομένως εκτός εθούσης. Αυτό ισχύει και για όσους συζητούν στο βάθος της εθούσης. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω να τελειώσουν αυτές οι συζητήσεις διότι μπορούν να διεξαχθούν και εκτός εθούσης. διότι τώρα έχουμε τη συζήτηση με την Τσεχική Προεδρία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ τον πρεσβευτή Ιβο Σράμεκ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλείας και Αμήνης και τον καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και τον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία την οποία ε, ε, είχαμε ε, στην υποαπιτροπή μας στα πλαίσια της στην αρχή της Τσεχικής Προεδρίας είχαμε σοβαρές ε, κρίσεις. Πρώτον η κατάσταση στη Γάζα και δεύτερον το θέμα της παροχής ε, φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αυτά τα θέματα εξετάστηκαν ή στην Επιτροπή Αμήνης και Ασφαλείας και υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες πρέπει επίσης να εξετάζονται. Σκέφτομαι το κοσφοπέδιο με την ε, αποστολή Όιλεξ για τη γεωργία με τους παρατηρητές και ε, με την ΕΣΑΤ ε, όπου αλλάζει η Προεδρία και θα ήθελα να, να ξέρω τι θα γίνει σε αυτά τα πλαίσια ε, πιστεύω ότι η πειρατεία είναι επίσης πολύ βασικό θέμα που μας απασχολεί και αρχή Ιανουαρίου μία ε, αποστολή του Κοινοβουλίου πήγε εις ε, την Αταλάντα διαπίστωσε η κατάσταση πάει καλώς συνάντησε τον Άβαρχο Τζόνς και ελπίζω ότι στις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσει και αυτός να επιστρεφεί την Επιτροπή μας. Άλλα θέματα μας απασχολούν επίσης. Η δυνάμεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από την Γαλλική Προεδρία ιδίως όσον αφορά την, σχετικά με την πολιτική άμυνα και την στρατιωτική άμυνα και αναρωτιέμαι τι πρόκειται να γίνει με τους 60.000 αυτούς στρατιώτες. Αυτοί έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν ομάδες ε, μαχής, υπάρχουν ομάδες τσέχων και Σλοβάκων που πρέπει να λάβουν θέση ως ο νουπο και θα ξέρω, ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις ομάδες και επίσης ε, ότι δεν θα πρέπει ε, η Προεδρία μόνο να ασχολείται με τον, ε, την ε, με τον προγραμματισμό αλλά και με τη διεξαγωγή ε, των ε, δράσεων και θα ήθελα να ξέρω πώς θα λύσετε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την Τουρκία το οποίο χρειάζεται, δυσχεραίνει την εφαρμογή του προγράμματος Βερολίνο ΣΥΝ. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο και ελπίζω ότι θα μας απαντήσετε σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχατε απόλυτο δίκιο. Το πρόγραμμα για ορισμένες προτεραιότητες ε, καταρτίστηκε και χρειάστηκε να εφαρμοστεί ε, με την ε, πρώτη μέρα της Προεδρίας μας διότι υπήρχε η κρίση σχετικά με το φυσικό αέριο τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και πολύ χρόνος χρειάστηκε να ε, καταναλωθεί για να επιληθούν ουσιαστικά αυτές οι δύο κύριες κρίσεις. Ε, εμείς ασχοληθήκαμε ε, ιδίως με την Μέση Ανατολή και η Τσεχική Προεδρία ήταν πολύ ενεργή στο θέμα αυτό οργάνωσε ε, επισκέψεις της Τρόικα ήδη από τις πρώτες ημέρες του έτους 2009 ο κύριος Σβάρτσεμπεργκ με τον Χαβιέ Σολάνα και την Επίτροπο Φερέρο Βάλτνερ πήγαν στην ε, ε, Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στα Παλαιστινιακά εδάφη κατά τρόπον ώστε να προσπαθήσουν να επιλύσουν την, ε, κράτη, την κρίση και να ε, προσπαθήσουν να ε, προωθήσουν τις προσπάθειες και στη συνέχεια σε επαφή με τους πρωθυπουργούς των κρατών της περιοχής και ε, ουσιαστικά συζητήσαμε πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τη εξέβρεση μίας λύσης. Δύο θέματα ουσιαστικά συζητήσαμε. Τα, βεβαίως τα θέματα ήταν πολλά, αλλά τα βραχυπρόθεσμα θέματα που συζητήσαμε καταρχήν ήταν ε, η ανθρωπιστική δράση, τι μπορούσε να γίνει και τι ζητούμε από τους Ισραηλινούς για να μπορέσουμε να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια και δεύτερον σχετικά με τις ανησυχίες των Ισραηλιών για την ασφάλειά τους λόγω του λαθρεμπορίου ε, πολεμοφοδίων και όπλων στη Γάζα. Αυτά ήταν τα ουσιαστικά θέματα που συζητήσαμε. και εφαρμόσαμε αμέσω το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, για βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη δράση. Όπως σας είπα, ε, καταρχήν ε, ανθρωπιστική δράση και αποφυγή λαθρεμπορίου όπλων και πολεμοφοδίων αναπτύξαμε ορισμένες ιδέες σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτά τα πλαίσια και ζητήσαμε να παραμείνουν ανοιχτά τα σημεία διελεύσεως μιλούμε για την ανοικοδόμηση την ενδοπαλαισθηνιακή συμφιλίωση που είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για οποιαδήποτε μελλοντική λύση ειρήνης και την, ε, την επανάληψη της ειρηνιστικής διαδικασίας. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία του καταλόγου τα οποία συζητούνται και συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε. Ο Χαβιλέ Σολάνα είναι αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και συζητάμε τους ομολόγους του και ο Λουί Μισελ, ε, συζητάμε τους ε, Αιγυπτίους και τους Ισραηλινούς και θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας στα πλαίσια αυτά. Επίσης ε, μας ενδιαφέρει η βραχυπρόθεσμη σκοπιά, δηλαδή τι μπορεί να γίνει αμέσως όπως προανέφερα, αλλά ακόμη και αυτά είναι δύσκολα πράγματα, διότι ε, θα πρέπει να έχουμε ένα ομόλογο από την άλλη πλευρά και ε, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής μεταξύ της Φατάχ και της Αμάς και προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση και οι ε, Αιγύπτιοι έχουν εμπλακεί ενεργά στο θέμα αυτό όπως άλλωστε και η Παλαιστίνη της Δυτικής Όχθης και έχουν παρουσιάσει τις ε, δυνάμεις της ε, ε, δυτικής όχθης για να μπορούν να παρίστανται. Ε, αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες συνεχίζονται και ε, ζητούμε βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να στείλει αμέσως ε, δυνάμεις ε, μόλις ε, θα έχει και την εξουσιοδότηση των Ισραηλινών. Όσον αφορά τις αποστολές αστυνόμευσης στο Ιούπολ Θα σας έλεγα ότι η αποστολή αυτή έχει ενισχυθεί παρόλη τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί και αναπτύσσουμε δραστηριότητες στο θέμα της καταπολέμησης της εγκληματικότητος και της προσαγωγής στη δικαιοσύνη. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και εκεί. και ζητούμε επίσης σύνδρομη για να ενισχυθεί η αποστολή μας. Αναφέρατε επίσης, δεν ξέρω αν θα καλέψω όλα τα θέματα ή να αναφέρω μόνο ορισμένα, Μπορείτε να παρουσιάσετε μία σύντομη γενική επισκόπηση και μετά θα υπάρξουν και ερωτήσεις. Αναφέρατε επίσης την Αταλάντα. σαν ένα θέμα που απασχολεί την Επιτροπή και θα σας έλεγα ότι ήταν ε, η πρώτη ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη επιχείρηση ε, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της πειρατείας ε, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα αυτό είναι μακροπρόθεσμα και η λύση δεν θα εξευρεθεί στη θάλασσα αλλά στην ξηρά γιατί πρόκειται μάλλον για συμπτώματα και όχι για την ουσιαστική αιτία αλλά δεν έχουμε άλλη εναλλαγή διότι τώρα πρέπει ε, ε, λόγω του, της εκτάσεως του προβλήματος ε, να επέμβουμε στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες επηρεάζονται. Η επιχείρησή μας ξεκινά από τη Βορεία Οδό και προβλέπουμε ότι θα διατηρηθεί επί ένα έτος. Έχουμε καλέσει και άλλα να συμμετάσχουν και μεταξύ αυτών των χωρών είναι η ε, Ελβετία, η Κροατία, η Ουκρανία οι οποίες εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να συμβάλλουν στην Αταλάντα. Ε, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες έχουν αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή. Μέχρι στιγμής η, ε, η ναυτική αυτή δύναμη αποτελείται από τέσσερις φρεγάτες, μία ελληνική, μία γερμανική, μία γαλλική ε, και ε, υπάρχουν και ελικόπτερα και, και αεροπλάνα ειδικά σε προθαλασσώσεις υπάρχουν και τρία σουηδικά πλοία τα οποία θα προσθεσούν ίσως το καλοκαίρι καθώς επίσης και μία φρεγάτα ακόμη. Η εντολή της αποστολής ε, τη βασική, ο βασικός της στόχος είναι η προστασία της ναυτιλίας για το παγκόσμιο επιστημικό πρόγραμμα ε, και η ε, ασφαλής πρόσβαση εις τον Περσικό κόλπο αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εντολή για να αποβιβαστεί στην ξηρά και ίσως το πιο δύσκολο ή μάλλον το πιο σημαντικό σημείο της προσπάθειάς μας είναι να συντονίσουμε τα πάντα, με ε, την ε, Αμερικανική δύναμη η οποία καθώς επίσης και τους Ρώσους να ε, συντονίσουμε δηλαδή όλες αυτές τις προσπάθειες στην περιοχή. Ίσως θα σας ενδιέφερε επίσης με τι, να γνωρίζετε τι γίνεται στη Βοσνία διότι έχουμε ένα φύλλο πορείας που είναι κάπως περίπλοκο για να εφαρμοστεί διότι ε, άλλαξε ο Σλοβάκος Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Σάλατσεκ έχει αντικαθασταθεί από κάποιον άλλον και ε, δεν ξέρουμε ε, αν θα χρειαστεί ε, αν θα χρειαστεί ένα νέο γραφείο ή ένα νέο άτομο υπάρχει εν πάση περιπτώσει ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε θα γίνει ένα ε, συμβούλιο για την εφαρμογή του προγράμματος το Μάρτιο για να δούμε αν το γραφείο αυτό θα αλλάξει μορφή και θα εξαρτηθεί κατά πολύ το μέλλον της αποστολής από τις αλλαγές στο γραφείο αυτή. Αν όμως όλα πάνε καλά Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μία μείωση της αποστολής και ε, η μη εκτέλεση της εντολής σημαίνει ότι θα καταρτηθεί μία δύναμη η οποία θα στηλίξει τις ε, ντόπιε ε, δυνάμεις Χρειαζόμαστε λοιπόν ακόμη μια εκτελεστική εντολή γιατί δεν θέλουμε να περιπλέξουμε την ε, πολιτική κατάσταση. Η κατάσταση ασφαλείας είναι αρκετά ήρεμη. Όπως είπαμε λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά είναι ένα πακέτο που μπορεί να οδηγήσουν σε, πιο, μια πιο σαφή εντολή και θα προσπαθήσουμε ε, ε, η εντολή η οποία θα ανανεωθεί να είναι μη εκτελεστική. Μια άλλη σημαντική αποστολή που θα έπρεπε να αναφέρω είναι το Αφγανιστάν. Ίσως έχετε ακούσει ότι ε, ενισχύουμε κατά πολύ την αποστολή μας εκεί η οποία πηγαίνει αρκετά καλά αλλά υπάρχουν βασικά θέματα ακόμη σχετικά με ε, τον συντονισμό και νομίζω το πολύ κανό νέο είναι ότι ε, έρχεται ένας ε, νέος ε, υπουργός, ο Αντβάρ, και το πιο βασικό θα είναι εις το Αφγανιστάν να προετοιμάσουμε τις εκλογές και να εξασφαλίσουμε ότι η αποστολή παρακολουθήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι ασφαλής. και να, ότι θα υπάρξουν ελεύθερες εκλογές. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Και τώρα ξεκινούμε τις ερωτήσεις. Έχουμε μία ερώτηση σχετικά με την Γάζα και το άνοιγμα των ε, συνόρων. Ποια είναι τα τελευταία νέα. Ε, οι, οι ε, επιθέσεις έχουν σταματήσει όσον αφορά τους πυλάβλους από τη Γάζα. Έχουν όντως σταματήσει. Και δεύτερον, Πώς αντιμετωπίζετε το λαθρεμπόριο όπλων μέσω των τούνελ και αυτό θα μπορέσει να, ε, να εξασφαλιστεί. Επίσης πιστεύετε ότι θα χρειαστεί ναυτικές δυνάμεις, πλοία ή διαφορετικά πώς θα παρακολουθεί κανείς ε, τα σύνορα αυτά και πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Ίσως μπορούμε να συγκεντρώσουμε διάφορες ερωτήσεις. Η κυρία έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να, πω να σχολιάσω δύο θέματα, αφενός το, τη Γάζα και αφετέρου το Αφγανιστάν. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει ε, να δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση διασυνοριακή ε, για τα ε, γεγονότα αλλά υπάρχει μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και ε, το Ισραήλ αρνείται να επιτρέψει να υπάρξει ε, παράδοση βοηθείας στην περιοχή. Ξέρετε ότι είναι δυνατόν να διέλθουν άτομα από τα σύνορα αλλά δεν είναι δυνατόν να μεταφέρει κανείς σε φορτηγά αυτοκίνητα με ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να παραμείνουμε απλοί παρατηρητές που δεν θα σχολιάζουν ε, όταν ε, το Ισραήλ αρνείται αυτά τα οποία έχει προσυπογράψει. Επίσης Όσον αφορά ε, τη στρατηγική η οποία ε, ε, αλλάζει σχετικά με την αλλαγή Προέδρου στην ευρωπαϊκή στις Ηνωμένες ε, Πολλές φορές έχουμε συζητήσει τα κριτήρια επεμβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αντιλαμβάνουμε ότι τώρα ο επικεφ επικεφαλής του ΝΑΤΟ έχει διατάξει παράνομες θανατώσεις ατόμων ε, και ε, ο, στρατηγός του ΝΑΤΟ αρνήθηκε να προβεί σε τέτοιες πράξεις στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρώπη έχει σχετικά με το θέμα αυτό μία κοινή θέση ή αν πρόκειται να έχουμε νέες ε, αμφισβητήσεις σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Αντιλαμβάνουμε αυτά τα οποία λέει ο συνάδελφός μου για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Παλαιστίνη και την κατάσταση στη Γάζα ειδικώ. Εσείς αναφέρατε ότι ε, ε, σας ανησυχεί η, ε, ότι θέλετε να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ αλλά τι γίνεται σχετικά με το, την άλλη πλευρά διότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα ελέγχθη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ε, την ε, εξέταση των εγκλημάτων πολέμου ε, και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και στις ευθύνες του Χαμάς έχει συζητήσει στο Συμβούλιο το θέμα του να θεωρεί στο Συμβούλιο τη θέση του της άμεσης διαπραγμάτευσης με το Χαμάς και θέλει να αλλάξει η ευρωπαϊκή θέση σχετικά με την Χαμάς. Και ε, ε, όταν, ε, όταν είχαμε ε, συζητήσει εις ε, το παρελθόν είχα ακούσει ότι μία εκπρόσωπος ήταν έτοιμη να μιλήσει με το Χαμάς την επομένη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες και των δύο πλευρών και ο γερουσιαστής Μίτσελ που εστάλθη από τον ε, πρόεδρο Μπάμε. Ξέρουμε αν θα υπάρξει επαφή με τον ε, γερουσιαστή Μίτσελ από τις πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Αταλάντα. Είπατε ότι ε, έχετε θέσει όρια σχετικά με την μακροπρόθεσμη επιχείρηση γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να επιτύχει και δεν μπορεί το πρόβλημα να λυθεί εάν δεν λυθεί το πρόβλημα ή στην ξηρά και όχι μόνο στη θάλασσα που αντιμετωπίζεται διότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει γίνει σχετικά με ε, την ε, επίλυση της καταστάσεως στη Σομαλία η οποία οδηγεί οδηγεί εις ε, την ε, ε, πειρατεία, στις πράξεις αυτές πειρατείες. Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει νόημα ιδίω τώρα με την αλλαγή πορείας και διαθέσεως Ηνωμένες Πολιτείας. Ε, διότι εκεί που η προηγούμενη διοίκηση των ΗΠΑ ε, ήταν πιεστική ε, τώρα βλέπουμε ότι αποσύρονται οι ακραίες δυνάμεις οι οποίες ήταν στην αρχή ε, σχετικά με, τον, με το Αφγανιστάν έχετε επαφές με τον κύριο Χόλμπρουκ ο οποίος έχει οριστεί από τον κύριο Ομπάμα για να ηγηθεί της αμερικανικής στρατηγικής για να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε ε, να κάνουμε θετικές κινήσεις στο Αφγανιστάν. Και τέλος σχετικά με τον Γουαντάναμο το οποίο αναφέρθηκε σχετικά με τις διατυπώσεις ασφαλείας που θα χρειαστούν σε ορισμένα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να δεχθούν ορισμένα από τα άτομα τα οποία κρατούνται έχοντας απαλλαχθεί από υποψίες εκ μέρους των Αμερικανικών αρχών. Μπορείτε να μας πείτε τι συζητιέται και αν υπάρχει στήριξη ε, για ε, δράση στο γεύμα αυτό που έγινε σε επίπεδο υπουργών ώστε να υπάρξει κάποια ε, οικονομική βοήθεια για την στήριξη των κινήσεων αυτών. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις, οπότε κύριε Πρέσβη έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με τις ερωτήσει Με τα προβλήματα του λαθρεμπορίου στη Γάζα και έχω να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα από ό,τι βλέπουμε από την ανάλυση Τα όπλα αυτά περνάνε μέσω της Σιναή από τα τούνελ αυτά, στην, από το ΣΥΝΕ, συγγνώμη, από τα ε, τούνελ αυτά στην Γάζα. Όταν μιλάμε λοιπόν ε, για ε, ναυτική πτυχή, είναι, αναφερόμαστε εδώ στην Ερυθρά θάλασσα. Γιατί κατά τα άλλα για να μην περάει τίποτα. Υπάρχει με αυτό τον ε, ε, τούνελ και οπωσδήποτε και των διοδίων, ε, των σημείων διόδου δηλαδή, γιατί αν υπάρχουν αυτά πάντα υπάρχει και κάποιο λαθρεμπόριο. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι να δώσουμε στους Αιγυπτίους κάποια τεχνολογία που θα τους επιτρέπει να βρούνε αυτά τα τούνελ. Φαίνεται υπάρχουν εκατοντάδες. Πολλά καταστράφηκαν, αλλά ακόμα πιο πολλά εξακολουθούν να είναι λειτουργικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τους Ισραηλινούς για να μπορέσει έτσι να διατηρηθεί η κατάβαυση του πυρός. Όσον αφορά τους πυράβλους στους οποίους αναφερθήκατε, φαίνεται ότι η εκεχηρία παραμένει. Οι Ισραηλοί είπαν ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της δικής μας επίσκεψης εκεί και της επίσκεψής τους εδώ ότι δεν θέλουν να καταστρέψουν τη Χαμάς αλλά απλώς να την αποτρέψουν από την ε, Όπω ε, πυράβλων. Όσον αφορά τις ερωτήσεις της Μπέρ, θα ήθελα να σας πω ότι τα να ανοίξουν τα σημεία αυτά διέλευση των συνόρων Εμείς βέβαια συζητάμε για το να ανοίξουμε το σημείο διέλευση ράφα, αλλά υπάρχει πρόθεση να διευρυνθεί βέβαια η προσπάθεια αυτή όταν οι προϋποθέσεις είναι κατάλληλες. και όλοι οι ενδιαφερόμενοι Ισραηλοί, οι Αιγύπτιοι εμείς και οι Παλαιστινιακές αρχές συζητούν το θέμα αυτό. Και ξέρουμε βέβαια πόσο πήγον είναι το θέμα και πόσο γλίγορα πρέπει να ολοκληρωθεί. Αναφέρατε επίσης ότι η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί δεν είναι επαρκής. πολλά κράτη-μέλη ζητήθηκε να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ και να βελτιώσουν την κατάσταση που υπάρχει. Και ο υπουργό μα ε, είναι σε επαφή με την Ελληνική και με τους πρέσβεις στην Ιερουσαλήμ και έχουμε την εντύπωση ότι βελτιώνει την κατάσταση. concerning uh, concerning the drug barons and in Afghanistan. Όσον αφορά το θέμα του Αφγανιστάν, και το θέμα των δολοφονιών εκεί. Πρώτη φορά το άκουσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε δεν προβλέπει κάτι. Ούτε άκουσα και το ΝΑΤΟ να προετοιμάζει κάτι. Ξέρουμε βέβαια ότι η κατάσταση είναι αρκετά πολύπλοκη. Και γι' αυτό θεωρούμε και τις εκλογές όσο σημαντικέ. Γιατί το επίπεδο διαφθοράς εκεί σε πολλούς τομείς της ε, αφγανικής ε, κοινωνίας είναι πάρα πολύ ψηλό. Uh, uh, Όσον αφορά το ε, έντυπα της κυρίας Κομές και την ερώτησή της για την ασφάλεια του Ισραήλ και τις ενισχύσει ασφάλειας των Παλαιστινίων ξεκίνησε από το ότι η Χαμάς δεν τήρησε τον κατάπαυση του πυρός και εξαπέλυσε πυράβλος στο έδαφος του Ισραήλ. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η κατάπαυση του πυρός να συνεχίσει και μετά να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Φυσικά οι Παλαιστίνοι έχουν εύλογες ε, ανησυχίε όσον αφορά την ασφάλεια, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί σαν τμήμα της ειρηνευτικής διαδικασία στην Ανάπολη, Όπω λέγεται, κάτω από την συλλογική αυτή προσπάθεια και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή η έφυγε. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναρχίσουμε μέσα στα πλαίσια της νέας κυβέρνησης. concerning the EU support for... Όσον αφορά την ε, ε έρευνα των ε, εγκλημάτων πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια το υποστηρίζει αυτό και υποστηρίζουμε και το ε, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που ζήτησε να γίνει η έρευνα αυτή. Και όπως είπατε και εσείς αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε μια Ισραηλινή έρευνα, γιατί το Ισραήλ είναι βέβαια μια δημοκρατική χώρα. Είναι ένα κράτος δικαίου, έχει κυβέρνηση και γι' αυτό πλήρως πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή Αν όχι θα το εξετάσουμε από κοντά και θα δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Η Χαμάς βέβαια είναι πιο μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα ερευνηθεί εκεί, ποιος θα το ερευνήσει, τι θα γίνει με τα εκεί εγκλήματα πολέμου. Ε, concerning, concerning... Όσον αφορά τον γερουσιαστή Μίτσελ. Ο Σολάνα το συνάντησε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτή, αλλά γενικά έχω να πω ότι σκοπεύουμε να έχουμε αυτές τις ε, επαφές με την νέα κυβέρνηση στις αρχές ε, του επόμενου μήνα. Θέλουμε να εξετάσουμε όλα τα θέματα. Ε, μέχρι στιγμής βέβαια δεν προλάβαμε, δεν υπήρχε αρκετό χρόνος και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να τα μελετήσουμε αυτά τα θέματα και να διαβουλευτούμε πάνω σε αυτά. Αταλάντα. Ναι, ξέρουμε βέβαια ότι δεν μπορεί να είναι επιτυχής η εξατία αυτή αν δεν λυθεί η κατάσταση στην Σομαλία. Το Ηνωμένα Έθνη βέβαια είναι η καλύτερη οργάνωση για να επιλύσει τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει ιδιαίτερο ενθουσιασμό από πλευρά τη Αφρικανική Ένωση να στείλουν στρατεύματα στη Σομαλία. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια που εξετάζεται στα Ηνωμένα Έθνη και εκεί είναι καλύτερο να εξεταστεί. Γιατί εμείς απλώς ε, τα συμπτώματα προσπαθούμε να κουράρουμε. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η αδυναμία της σημερινής μας πολιτικής. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενθουσιασμό για να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σομαλία. E e Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά υποστηρίζει ΝΕΜΣΑΜ και υποστηρίζουμε και την Αφρικανική Ένωση. διαθέτοντάς ό,τι δυναμικό και δυνατότητες έχουμε στην Σομαλία. και οπωσδήποτε είναι ένα καυτό θέμα για μας η Σομαλία παρόλο που θα έλεγα ότι είναι θέμα που αφορά την Αταλάντα. Και αυτό που είπα προηγουμένως για τις ε, επαφές μας στις Ηνωμένες αφορά τις ε, επαφές μας και για την Σομαλία με την κυβέρνηση. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Το ίδιο θα μπορούμε να πούμε για τον Ολμπρουκ και την ε, πολιτική τον είπα για το Αφγανιστάν. Αυτά όλα θα εξεταστούν σε συναντήσεις αρχές Φεβρουαρίου με τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γκοντάναμο. Για πολλά κράτη-μέλη το Γκοντάναμο ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε στην τελευταία συνάντηση των Υπουργών και υπάρχει νομίζω συνένεση ότι θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. και ότι χρειαζόμαστε να έχουμε μια ενωμένη θέση για το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Οι διαπραγματεύσει μόνο άρχισαν, έχουμε το θέμα αυτό στην μέση μας διάταξη. Το... Την Παρασκευή, ο κ. Δεκιάρκοφ που ήταν εδώ παρόν προηγουμένως, θα μας ενημερώσει. Ό,τι φορά την γενική κατάσταση και τις επιπτώσεις, υποθέτω ότι θα προετοιμαστεί κάποιο έγγραφο των εναλλακτικών που θα μπορούν να ακολουθούν και βάσει του εγγράφου αυτού θα πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μεταξύ θα μελετήσουμε τις εναλλακτικές αυτές, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα αυτό για την ε, επόμενη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με την Χίλαρη Κλίντον το Φεβράριο. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέσβη. Θέλω να υποβάλω άλλη μια ερώτηση. όσον αφορά το θέμα της ομάδας αυτής της ε, τσεχικής-σλοβακικής ομάδας και η Αναγκόμπας έχει μου φαίνεται μία ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομη ερώτηση. Εν ώψη της απόφασης της χθες που πήρε η Ρωσία για να σταματήσουν την εγκατάσταση πυράβλων στο Καλίνιγκρατ και εν ώψη αυτών που ακούμε από τη ΣΥΠΑ όσον αφορά το ότι η ε, κυβέρνηση του Ομπάμα ξανεξετάζει το θέμα αυτό σε εγκατάσταση πυράβλων. Ποια είναι η δική σας άποψη στην ε, Τσεχία και στην ε, ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, δεν θα προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το θέμα της ομάδας αυτής ε, της ε, Battle Group ε, της ομάδας μάχης αυτή τη στιγμή προχωρεί και μπορεί να εγκατασταθεί. Είμαστε έτοιμοι. Για το δεύτερο ήμιση του 2009 βέβαια. Όσον αφορά τους πυράβλους στο Καλίνγκρατ, και την άμυνα, δηλαδή την πυραυλική άμυνα, δεν άλλαξε τίποτα από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα. Υπογράψαμε κάποιες συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ μέχρι στιγμής και είδαμε τι ελέγχθη από τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Αλλά πιστεύουμε ότι παρόλο που υπάρχουν κάποιες ιδέες σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή ρόλου όσον αφορά κάποιους πυράβλους μεσοβελληνικούς ή στρατηγικής. Δεν υπάρχει όμως τίποτα, τίποτα συγκεκριμένο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίσως κάποια πρώτα μηνύματα, αν θέλετε, ότι κάτι ίσως μελετάτε αλλά δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσει μεταξύ της δικής μου κυβέρνησης και της νέας ε, Αμερικανικής κυβέρνησης για ενδεχόμενες αλλαγές. Είναι, είναι βέβαια και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα συζητηθεί μεταξύ του Υπουργού με και της Υπουργού κυρίας Κλίντον. Δεν σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. και από πλευράς ε, Ρωσίας πρόκειται για μια χειρονομία. Ξέρω εγώ πώς να σας το αποκαλέσω. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίση ότι μέχρι στιγμή δεν είχαν εγκατασταθεί καθόλου πύραυλοι. Κανένα πύραυλο. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν το θέμα αυτό τη ε, ημερησία μου διαδέξη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη.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 ποιος θα, θα λάβει το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αναλαμβάνουμε ότι τώρα η Γάζα θα μιλήσει ε, ε, για τη Γάζα θα μιλήσουμε. Ποιος λοιπόν θα σχολιάσει σχετικά με τη Γάζα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Αψίδης από την Ρέλεξ F3. Κύριε Πρόεδρε, το όνομά μου είναι Αψίδης, είμαι στην ε, ε, Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή και ε, είμαι υπεύθυνο και για να παρουσιάσω την κατάσταση στη Γάζα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Ζων Κλοντ Βερό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της άλλης, της άλλης διευθύνσεως της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, η Γάζα είναι ε, το προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν είναι και ο μόνος υπεύθυνος ανά τον κόσμο. Ίσως θυμάστε ότι ήδη το Δεκέμβριο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπήρχε μία τριμερής επιτροπή της Προεδρίας ε, ε, που πήγε στην περιοχή, μετά πήγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά υπήρξαν συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητώντας ε, άμεση κατάπαυση του πυρός η οποία έγινε αποδεκτή μονομερός από κάθε πλευρά και είναι πολύ ευάλωτη διότι σύμφωνα με τα τελευταία νέα σήμερα το πρωί υπήρξαν δύο πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύθησαν και υπήρξε και απάντηση από τις Ισραηλινές ε, δυνάμεις άρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής. Έχουμε συνεχείς επαφής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις αρχές του Ισραήλ αλλά και σε συνεδριάσεις την προηγούμενη εβδομάδα με την ε, Υπουργό Εξωτερικών Λίβνη, ε, με τους Αιγυπτίους, Ιορδανούς και με το Υπουργείο Εξωτερικών ε, της Παλαιστίνης, ε, τους Τούρκους, είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Δευτέρα και έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης διότι πρέπει να δράσουμε και η πρώτη πρωτοβουλία και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προσφέρει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος για να μπορέσουμε να επιλύσουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός σε αυτό το θέμα. Πέραν της ανθρωπιστικής βοηθείας υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, τους οποίους θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε συγχρόνως. Ένα πολύ βασικό θέμα είναι το συνεχές ε, και ε, διαρκείας άνοιγμα των σημείων διελεύσεως αλλά και των άλλων σημείων που είναι σημαντικά αφενός για την, ε, ε, για την ε, προσφορά ανθρωπιστικών υλικών αλλά επίσης και άλλων στοιχείων που θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση στη συνέχεια. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η ε, αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, του λαθρεμπορίου όπλων, των δραστηριοτήτων που είναι πολύ σημαντικό σημείο για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το θέμα του να υπάρχει ένας ομόλογος στη Γάζα είναι πολύ βασικό και για τις δραστηριότητες τις ανθρωπιστικές και για την ανοικοδόμηση. Βέβαια υπάρχει ένας γενικός ε, υπεύθυνος ε, με την στήριξη του Μπάσκετ του Φαγιάντα δεν ε, υπάρχει η αρχή αυτή δεν, ε, δεν γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο και θα πρέπει να βρούμε ένα ομόλογο ο οποίος να είναι αποδεκτός και ε, στο τέλος της, του καταλόγου που πρέπει να είμαστε που να είμαστε ενεργοί ε, είναι το θέμα της, ε, ε, της προθήσεως της ειρηνευτικής διαδικασίας πράγμα το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος το οποίο θα μπορέσει να ζήσει δίπλα στο Ισραήλ ειρηνικά. Αυτή είναι η εισαγωγή μου κύριε Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας μαζί μαζί με τους συναδέλφους να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα και σε διευκρινήσεις ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες ε, τις οποίες έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σολάνα είναι στην ε, περιοχή για να ε, προωθήσει με τις Αιγυπτιακές και τις Ιταλικές αρχές τη την ε, εξασφάλιση της ε, ειρήνης και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια και να βοηθήσουμε τον Παλαιστινιακό λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην ε, Άννα Γκόμες. Καταρχήν δεν βλέπω να έχετε ερωτήσεις. Νόμιζα ότι τουλάχιστον μία θα είχατε. Οπότε τότε εγώ έχω μία ερώτηση σύμφωνα με τις πληροφορίες σας ποιες είναι οι πιο επίγουσες ανάγκες του πληθυσμού και ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε καταρτήσει. Ευχαριστώ. Σαφώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες και οι ανάγκες για μία σύντομη ανάκαμψη είναι βασικές. Τα σημεία διελεύσεως είναι ανοιχτά αλλά όχι συνεχώς. Κατόπιν ε, των, ε, των ε, γεγονότων των προχθεσινών εχθές έκλεισαν. Τα σημεία αυτά πρέπει να είναι ανοιχτά και να μένουν συνεχώς ανοιχτά διότι οι ποσότητες των ανθρωπιστικών αγαθών που φτάνουν είναι ανεπαρκείς. Μόνο 200 φορτηγά μπορούν να περάσουν τώρα ενώ προηγουμένως πριν από τον αποκλεισμό γνωρίζαμε ότι χρειαζόντουσαν 500 με 600 φορτηγά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο τελευταίο έτος, ιδίως μετά, ε, πριν από την ε, ε, τον κρίση οι ανάγκες για ανθρωπιστικά αγαθά αλλά και για αγαθά όπως σωλήνες, τσιμέντο, οικοδομικά υλικά που χρειάζονται ε, για να μπορέσει να αποκατασταθεί το δίκτυο ηλεκτρισμού και νερού που κατεστράφει χρειάζονται και ε, υπάρχουν πάρα πολλά σε εκατοντάδες ατόμων των οποίων η οικονομία καταστράφηκε που τώρα ε, εξαρτώνται από την εξωτερική βοήθεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι ποσότητες έχουν αυξηθεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρώτον πρέπει να υπάρχει άμεση, ε, ε, άμεσο άνοιγμα όλων των σημείων διελεύσεως και δεύτερον να γνωρίζουμε τι ποσότητες χρειάζονται. Επίσης πρέπει να δούμε το είδος των αγαθών που χρειάζονται διότι υπάρχουν ε, διαφορές όσον αφορά τα ανθρωπιστικά υλικά που χρειάζονται διότι για μας δεν πρόκειται μόνο ε, για τρόφιμα και φάρμακα αλλά και ε, άλλα υλικά που χρειάζονται για μία σύντομη ανάκαμψη και για να γίνουν και οι επισκευές. Ε, χρειάζεται το προσωπικό, το ανθρωπιστικό να έχει πλήρη πρόσβαση και τώρα υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχουν καθυστερήσεις στη χορήγηση αδειών οπότε όντως θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση του προσωπικού και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, πράγμα το οποίο είναι βασικό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχει και μία άλλη πολύ σημαντική ανάγκη κάποιου στοιχείου το οποίο δεν είναι ίσως προφανές, ε, μετρητά. μετρητά. Αυτό που δεν υπάρχει είναι χρήματα, μετρητά. Διότι έχει καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και οι Ισραηλινές αρχές για να αποφύγουν ροές ε, χρηματοδοτήσεως προς το Χαμάς έχουν περιορίσει την πρόσβαση μετρητών και μετά από πολλά διαβήματα ε, επέτρεψαν την, ε, την διέλευση των μισθών για το προσωπικό της Ούνρα. Αλλά αυτό δεν επαρκεί οι ε, διάφοροι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, η βοήθειά μας η ίδια υποβιβάζεται και μειώνεται διότι δεν είναι δυνατόν μέσω του μηχανισμού μας να χρηματοδοτήσουμε τα άτομα τα οποία χρειάζονται μετρητά και η οικονομία δεν μπορεί να συνέλθει. Ίσως ο συνάδελφός μου, ο Ζων Κλοντ, θα έχει κάτι περαιτέρω να πει σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω τις βασικές αρχές που έχουν, τα, βασικά σημεία που έχουν ε, διαπιστώσει. Καταρχήν, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως ε, για τους άμαχους ε, που δεν μπόρεσαν να γυρίσουν σπίτια τους. Χρειάζεται επίσης βοήθεια ούτως ώστε να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι Επίσης είναι πολύ σημαντική η παροχή νερού. Μετά από 18 μήνες μπλόκου ήδη υπήρχε πρόβλημα με την παροχή νερού διότι δεν περνούσαν τα ανταλλακτικά για να αποκατασταθεί το για να αποκατασταθούν οι σωληνώσεις του νερού Και σήμερα μετά τους βομβαρδισμούς οι Ισραηλινοί πάλι έχουν επιφυλάξει στο να αφήσουν να μπουν σωλήνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους. Πρόκειται όμως για μια απόλυτη ανάγκη. Η βενζίνη επίσης Και υπάρχει φυσικά και το πρόβλημα των ελαχίστων φορτηγών που μπορούν να μπουν στη ζώνη της Γάζας. Πέρυσι είχαμε, 73, είχαμε δεσμεύσει 73 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ακόμη ξοδεύονται. Με το 9 Ιανουαρίου είχαμε δώσει ένα συμπλήρωμα Και έχουμε δηλαδή 58 εκατομμύρια ευρώ όπως ανήγγειλε ο Λουί Μισελ και τα 32 πάνε στη Γάζα. Βέβαια ακόμη οι ανάγκες δεν έχουν αξιολογηθεί γιατί η αρμόδια αποστολή του ΟΗΕ είναι αυτή που κάνει τις αποτιμήσεις και τις εκτιμήσεις και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν και τις δυνατότητες πρόσβασης που θα έχουμε θα κανονίσουμε τη βοήθεια. Για τις αποζημιώσεις τώρα. Έχουμε πραγματικά βάσιμη αξιολόγηση του τι έγινε. Έχουμε στοιχεία σωστά. Και εκτός αυτού υπάρχει πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες από τον για να γίνει η αξιολόγηση αυτή. Και δεύτερον, όσον αφορά αυτήν την αποστολή των Αμναφά, Εγώ είδα τέτοιες αποστολές στις οποίες είχε εμπλακεί έντονα η Κομισιόν τώρα αυτή η αποστολή στην Ράφα όταν αναζωογονηθεί θα υπάρχει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά ποιον τρόπο. Euh, Σχετικά με τις εκτιμήσεις γίνονται από αυτούς ε, που ήταν παρόντες πριν από τον πόλεμο. Και το ΣΕΣΕ που ήταν φυσικά επιτόπου που θα γίνουν δηλαδή και θα γίνουν και οι εκτιμήσεις ε, των σπιτιών που γκρεμίστηκαν ή των μερικά καταστραμμένων σπιτιών Ανέφερα βέβαια αυτά τα... Ανέφερα δύο μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά υπάρχουν και άλλες που, υπάρχουν, που είναι στην περιοχή και οι οποίες ανταποκρίνονται τα, το μάξιμουμ δυνατόν. Εμείς βέβαια ε, δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες τις οποίες έχει η Κομισιόν. Να συμπληρώσω κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα της ΡΑΦΑ υπάρχει και μία αξιολόγηση των ε, άμεσων αναγκών. Εξετάζουμε στη Γάζα ήδη αυτό το θέμα ιδίως εκεί που υπάρχουν ε, κάποιες ε, κάποιοι εξοπλισμοί που δεν έχουν εκραγεί ή και όσον αφορά την ε, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη του πληθυσμού. Το 50% του πληθυσμού εκεί είναι παιδιά 115. 15. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ έντονες τραυματικές επιπτώσεις της ε, ε, σύραξης στα παιδιά. Εξετάζουμε την κατάσταση αυτή και εξετάζουμε και το μέσο σταθερότητας που προβλέπει κάποιος ελέγχους. Όσον αφορά το θέμα της ε, ε, αποστολής στη Ράφα, κινητοποιούμεθα, ξέρετε ότι το ο προσωπικό περιμένει, είναι έτοιμο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι όροι της σταθερότητας, να υπάρχει συμφωνία όλων των συμμετεχόντων. Ε, η Κομισιόν είναι έτοιμη, συμμετείχαμε και περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης των ζημιών όσον αφορά το σημείο διέλευσης της ράφα που πυροβολήθηκε λίγο πριν από την ε, ε, του πυρός. Θα πρέπει να δούμε εάν επλήγει, ποιε είναι οι βλάβες και ως Κομισιόν οπωσδήποτε είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε περαιτέρω αποστολές, αν υπάρχουν κάποιες, ή αν υπάρχει μια διαφοροποίηση ή διεύρυνση της, απο... της εντολής. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, αναφέρθηκα σημασία των σημείων διεύλευσης όχι μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και για εμπορικούς λόγους και για τους ανθρώπους τους ίδιους και υπάρχει δυνατότητα ορισμένα από αυτά τα σημεία διαρρεύσης, όχι μόνο τη Ράφα, αλλά και άλλα, εκείνα που περνάνε από τη Γάζα στο Ισραήλ και αντίστροφα, να βελτιωθούν στην ποιότητά τους. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να επανέλθουμε στο τάτους κβό και μια κατάσταση όπου υπάρχει ένα μπλοκάρισμα και της οικονομικής ζωής μετά από την πρώτη φάση της ε, οικονομικής ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας συγγνώμη, να περάσουμε σε μια οικονομική ε, ανάκαμψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, εσείς εξετάζετε το θέμα της αποστολή τη Ράφα και όχι μόνο αυτή αλλά και τα άλλα σημεία διάλευσης. Ναι, ναι, αυτή είναι η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου και οπωσδήποτε αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι από τα θέματα που θα συζητήσουν ο υπότος εκπρόσωπος σίγουρα αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις δεν βλέπω να υπάρχουν. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους παρόντες. Καλή συνεδρίαση.